Uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση. Το πρώτο μας θέμα είναι η παρουσίαση της Μαρή Τερέζ Σάντζε Σμιθ για την Ευρωπαϊκή ημέρα συνεργασίας ανταλλαγή απόψεων προβλέπεται με κάποιους συναδέλφους από την Interact και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρέπει να ξεκινήσουμε, ξέρετε, γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Μαρή Τερέζα, έχει το λόγο. Euh, Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους. Χαίρομαι ιδιαίτερα που μπορούμε σήμερα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχουμε αυτή την παρουσίαση για τις ημέρες Ευρωπαϊκής Συνεργασίας. Ευχαριστώ την Πρόεδρο και βεβαίως την Επιτροπή. Ξέρετε ότι προέρχομαι από μια τέτοια δεσυνοριακή περιοχή μεταξύ Γαλλίας και Ισπανίας και η συνεργασία αυτή είναι κάτι το οποίο με απασχολεί καθημερινά. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να δει κανεί την οικοδόμηση της Ευρώπης και η συνεργασία μεταξύ δύο περιοχών, μεταξύ δύο χωρών είναι εξαιρετικά σημαντική, ιδιαίτερα σήμερα που περνάμε αυτή την κρίση. Βλέπουμε ότι Σήμερα τα στατιστικά στοιχεία, οι δημοσκοπήσεις μας δείχνουν ότι υπάρχει μια εσωστρέφεια και μια αυτοπροστασία, κάτι το οποίο θα πρέπει να καταπολεμήσουμε. Η συνεργασία λοιπόν ξαναδίνει ένα νέο ευρωπαϊκό πνεύμα και θα πρέπει να ενισχύσουμε αυτή τη συνεργασία. Τα σύνορα αντιμετωπίζονται σαν διαχωριστικές γραμμές, σαν σημαίες έντασης. Αυτό θα πρέπει να το ξεπεράσουμε και αυτή η συνεργασία θα πρέπει να μας βοηθήσει να φτάσουμε σε περισσότερη, καλύτερη ανταγωνιστικότητα, να βελτιώσουμε την συνεργασία, τα πλεονεκτήματα των διαφόρων περιοχών που ουσιαστικά αλληλοσυμπληρώνουν τις περιοχές μας. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε νέες προσκλήσεις. Το 2011 η έκθεση της οποίας ήμουν ε, εισηγήτρια για το 2013 και το μέλλον αυτής της συνεργασίας, μας έδειξε ότι δεν υπάρχει αρκετή συνεργασία μεταξύ των περιοχών, ενώ η χρηματοδότηση είναι καλή. Βλέπουμε σήμερα ότι και οι πολίτες και οι διοικητικές ε, αρχές και οι φορείς δεν αντιμετωπίζουν σήμερα την εδαφική αυτή συνεργασία σαν ένα πλεονέκτημα. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσουμε μια μεγάλη εκστρατεία για να προωθήσουμε την συνεργασία κυρίως σε αυτές τις διασυνοριακές περιοχές. Για πρώτη φορά φέτος μετά από πολλούς μήνες συνεργασία αυτή η εκστρατεία θα ξεκινήσει χάρη στο Interact και τους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Πάνω από 70 προγράμματα σε πάνω από 40 χώρες ξεκίνησαν στις 21 Σεπτεμβρίου, σε αυτή την ημερίδα, με εκθέσεις, ε, με διοργανώσεις και με προγράμματα τα οποία φαντάζομαι ότι θα στεφθούν από πολύ πτυχία. στην περιοχή μου, στην ε, πόλη Παμπλούν. Ξεκίνησε μια διοργάνωση για να προωθήσει την διασυνοριακή συνεργασία. Πάνω λοιπόν από 70 προγράμματα, μεταξύ των οποίων και προγράμματα όπως αυτό προ... μας παρουσιάζει ο Ζων για τη Γαλλία και τη Βαλονία. Ο κύριος Μοντάν, ο οποίος είναι συντονιστής του προγράμματος Interactive Βιέννη, συμμετείχε στην οργάνωση αυτής της ημερίδας, την 21η Σεπτεμβρίου. Ξεκίνησε λοιπόν αυτή η ημερίδα με συμμετοχή του Επιτρόπου Ιωάννης Χάν, της ε, Προέδρου της Επιτροπής και της Ερικα Μάνερ, η οποία είναι συντονίστρια και θα ακολουθήσει ένα κοκτέιλ. Ξέρετε ότι πάντα μια τέτοια συνεργασία πρέπει να ξεκινήσει από μια τέτοια γιορτινή διοργάνωση. Θα ήθελα πριν δώσω το λόγο στον κύριο Μοντάν να ευχαριστήσω όλους όσους βοήθησαν στη διοργάνωση αυτή, η οποία κατά την άποψή μου θα βοηθήσει στο να γεφυρθεί το χάσμα μεταξύ των πολιτών της Ευρώπης. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μοντάν από το Interact έχει το λόγο. Um, I can't see On behalf of the Interact program, I would like to thank Mrs. Hübner, the chair of the... Εξ ονόματος uh, του Interact, θέλω να σε ευχαριστήσω κυρία Χιούμπνερ για την σημερινή σας πρόσκληση. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα θερμά την κυρία σας για την πρόσκληση του προγράμματος Interact να σας ενημερώσει για αυτή την Ευρωπαϊκή Εκστρατεία για την Ευρωπαϊκή Μέρα Συνεργασία. Είναι ε, μια πρωτοβουλία που θα λάβει χώρα αυτήν την εβδομάδα. Και θέλω να ευχαριστήσω για την εδαφική συνεργασία, ε, για τη στήριξη μάλλον στην εδαφική συνεργασία δεν είναι η πρώτη φορά που δείχνει τέτοιο ενδιαφέρον για την εδαφική συνεργασία. Πάντοτε έδειχνε αυτό το ενδιαφέρον καθ' ε, την ε, δραστηριότητα της ε, σε αυτή την Επιτροπή και γενικότερα την πολιτική της σταδιοδρομία. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης ε, τα μέλη της Επιτροπής ΡΕΚΙ για τη βοήθεια που δίνουν σε αυτό το τομέα. Ξέρετε ότι η εδαφική συνοχή δεν λαμβάνει το μεγαλύτερο όγκο χρημάτων από την πολιτική συνοχή, αλλά λαμβάνει ένα πολύ σημαντικό κονδύλι. Είναι πολύ σημαντικό ε, και είναι πολύ ενδιαφέρουσε και προκλητικέ, αν θέλετε, οι δραστηριότητε που είναι Το πρόγραμμα Interact, όπως γνωρίζετε, είναι ένα πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας. Το πρόγραμμα αυτό δεν χρηματοδοτεί project, αλλά υποστηρίζει γενικά τα προγράμματα εδαφικής συνεργασίας σε όλη την Ευρώπη. Και δεν μιλάμε απλά για εδαφική συνεργασία, αλλά έχουμε και ειδικά project, όπως είναι τα ε, προγράμματα γειτονίας, τα προγράμματα ENPI για την συνεργασία δηλαδή ε, με τις κοινωνικές χώρες της Ένωσης όπως και την συνεργασία με τις προενταξιακές χώρες, χώρες δηλαδή που κάποια στιγμή θα προσχωρήσουν στην Ένωση. Και όλες αυτές οι χώρες συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή ε, ημέρα συνεργασίας. ότι συνολικά μιλάμε για πάνω των 90 προγραμμάτων λαμβάνοντα υπόψη τα προγράμματα της γειτονία και της πρωτεξιακής συνεργασίας και μιλάμε για ενίσχυση σε όλους τους τομείς. Για παράδειγμα, ενίσχυση για την διαχείριση προγραμμάτων, όπως είναι η αξιολόγηση, αλλά πτυχές των προγραμμάτων. Έπειτα υποστήριξη για την οικονομική διαχείριση, για τον έλεγχο, για την επικοινωνία, όπως και για την προετοιμασία τους για τη μελλοντική προγραμματική περίοδο. Επ' αυτή την έννοια ίσως να λάβατε και να διαβάσατε 15 σημεία τα οποία προετοιμάσαμε για τους ενδιαφερόμενους φορείς εδαφικής συνεργασίας. Αυτά τα 15 σημεία είναι μία σύνοψη ε, του τι επιθυμούμε μέσω αυτών των προγραμμάτων της μελλοντική προγραμματικής περίοδου. Ελπίζω να διαβάσετε αυτό το έγγραφο. Η Ευρωπαϊκή Μέρα συνεργασίας είναι μία από τις δραστηριότητες ε, στο πλαίσιο ε, των δραστηριοτήτων επικοινωνίας μας ε, στην Interact. Στόχος αυτής της εκστρατείας είναι η εδαφική συνεργασία να γίνει πιο γνωστή, πιο ορατή στον πολίτη. Και θέλω να πω ότι η κυρία Σμιθ ειδικά στη σημερινή εποχή, ε, κατανοεί ακριβώς ότι θα πρέπει η συνεργασία που γίνεται ανάμεσα ευρωπαϊκές περιφέρειες να γίνει γνωστή και να έρθει πιο κοντά στον Ευρωπαίο πολίτη. Οπότε να γνωρίζει ο Ευρωπαίος πολίτης τι γίνεται και αυτό να επηρεάσει πιο πολύ την καθημερινότητά του. Για την εκστρατεία αυτή να πω εντάχει τώρα πώς έγιναν όλα αυτά. Πρέπει να πάω λιγάκι πίσω τον Απρίλιο του 2011, όταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε την έκθεση του στόχου 3 για την Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία, έκθεση της κυρίας Σάντσα Σμιτ, και ήταν σαφές αυτή την έκθεση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το πρόγραμμα Interact θα πρέπει να προάγουν τα επιτεύγματα ε, της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας ε, πιο ισχυρά στους πολίτες. Να βρούμε ένα κοινό λογότυπο, μια εκστρατεία ε, ενημέρωσης, ώστε να γίνουν πιο γνωστά στον πολίτη τα αποτελέσματα αυτής της δραστηριότητας. Ένα μήνα μετά την έγκριση της έκθεσης ξεκινήσαμε και εμείς τη δουλειά. Ξεκινήσαμε με λίγα, μια ομάδα προγραμμάτων, λάβαμε πολύ ισχυρή υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ευθύ εξ αρχή, αλλά και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχαμε ενθαρρυντικά λόγια και από τη δική σα Επιτροπή πιο συγκεκριμένα. Και σιγά σιγά, μέσα από τον άμεση χρόνο που πέρασε, λάβαμε όλο και πιο πολλές αιτήσει για την προσχώρηση σε αυτή την εκστρατεία ενημέρωση, όλο και πιο πολλά προγράμματα συμμετέχουν. Όπως ε, νωρίτερα είπε η κυρία Σάντσε Σμιθ, αυτή η εκστρατεία συνίσταται σε μία σειρά εκδηλώσεων που λαμβάνουν χώρα στις εγκαταστάσεις μας ή στις περιφέρειες εκείνες όπου δραστηριοποιούνται προγράμματα εδαφική συνεργασία αυτή τη στιγμή έχουμε 77 προγράμματα συγκεκριμένα. Δεν μιλάμε μόνο για προγράμματα εδαφική συνεργασία, αλλά και προγράμματα γειτονία και προτεξιακά προγράμματα. Και έχουμε πάνω από 100 εκδηλώσει όλη την Ευρώπη και πάνω από 40 συμμετέχουσε χώρε. Όλα λοιπόν αυτά τα προγράμματα και τους συμμετέχοντες ε, επιλέξαμε ότι η Ευρωπαϊκή ημέρα συνεργασία είναι η επόμενη Παρασκευή, 21 Σεπτεμβρίου, αλλά επειδή είναι πολλά τα προγράμματα, πολλοί είναι οι εμπλεκόμενοι, δώσαμε τη δυνατότητα οι εκδηλώσεις να είναι διάσπαρτες μέσα σε όλη την εβδομάδα. Οπότε θα ε, έχετε τοπίσει εκδηλώσεις και σήμερα και αύριο και την Παρασκευή βεβαίω. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από αυτό το αποτέλεσμα και από την επιτυχία της όλης εκστρατείας. Όπως θα βλέπετε και στις οθόνες σας, έχουμε δημιουργήσει ένα website. Το βλέπετε την ε, οθόνη. Ανοίγοντας λοιπόν αυτό το website θα βρείτε ένα χάρτη των εκδηλώσεων που λαμβάνουν χώρα σε όλη την Ευρώπη. Είμαι σίγουρη ότι εκδήλωση που είναι πιο κοντά στη δική σας περιφέρεια. Επίσης έχουμε σελίδα ε, και στο Facebook και στο Twitter λογαριασμό έχουμε και εκεί μπορείτε να μας παρακολουθήσετε πιο στενά και να δείτε πώς εξελίσσονται αυτές οι εκδηλώσεις. Επίσης έχουμε πολύ καλά παραδείγματα δραστηριοτήτων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορείτε να παρακολουθείτε μέσω του website μας. Πολύ διάφορες δραστηριότητες όπως ε, θεατρικά έργα. Διασυνοριακά ε, έχουμε πολύ ενδιαφέρουσες θετικές εκδηλώσεις α, στα σύνορα Κροατίας-Ουγγαρίας θεατρικά έργα που προσπαθούν να δημιουργήσουν μια εγρήγορση για τα θέματα των αρκοπεδίων. Επίσης, ε, έχουμε διοργανώσει έναν αγώνα δρόμου και αυτό γίνεται ανάμεσα στη Λετωνία και τις γειτονικές χώρες. Επίσης, υπάρχει μια πολύ καλή δραστηριότητα ανάμεσα στην Ελλάδα και την και Βλέπετε ότι ειδικά η θάλασσα που χωρίζει την Άρη και την Ιταλία θα τύχει πολλών εκδηλώσεων ε, και θα καλούμε λοιπόν να μπείτε στο website και να δείτε λεπτομέρειες. Επίσης δημιουργήσαμε και ένα βιντεάκι που κάνει την εκκίνηση της εκστρατείας. Θα το δούμε τώρα, δεν είναι μακρύ, είναι πάρα πολύ ωραίο βίντεο.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 Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πρόεδρος. Θα καλέσω τώρα τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Χιούγνερ. Εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα θέλαμε να σε ευχαριστήσουμε για την ευκαιρία που μας δίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παρουσιάσουμε και να λανσάρουμε αυτή την εκστρατεία προώθησης των προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Συνεργασίας, γνωστή πρωτοβουλία με την ονομασία Ευρωπαϊκή ημέρα Συνεργασίας. Γνωρίζουμε η πρόεδρος διακόπτει και λέει σε ισπανικά στον εκπρόσωπο της Επιτροπής να μιλάει πιο κοντά στο μικρόφωνο. Ναι, ναι. Θέλω πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω, λέει και πάλι ο μιλητής, για την πρόσκληση. Και δεύτερον, να επισημάνω τη δουλειά που έχει γίνει και ανταποκρίνεται στα αιτήματα της έκθεσης της κυρίας Σάνσε Σμιθ που κάποια χρονική στιγμή μίλησε για την έλλειψη προβολής και ορατότητας των αποτελεσμάτων που έχουμε επιτύχει μέσω των προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας. Ξεκινά λοιπόν σήμερα αυτή η ενημερωτική εκστρατεία ακριβώς για να δώσουμε μεγαλύτερη προβολή στα προγράμματά μας. Θεωρούμε επίσης ότι είναι μια σημαντική συγκυρία αυτή για την εδαφική συνεργασία, καθώς αυτή τη στιγμή που γίνονται διαπραγματεύσεις για την επόμενη προγραμματική περίοδο, η εδαφική συνεργασία που είναι ο δεύτερος στόχος της πολιτικής συνοχής, βλέπουμε πώς μπορεί πραγματικά η εδαφική συνεργασία να είναι παρούσα σε όλα τα προγράμματα πολιτικής συνοχής και όχι μόνο ε, στην, τη στενή έννοια της εδαφικής συνεργασίας. Έχουμε τώρα και ένα εργαλείο στα χέρια μας, έναν ειδικό κανονισμό που συζητήθηκε και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που θα ρυθμίσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και το τι ακριβώς μπορεί να προσφέρει στον ενδιαφερόμενους. Όπως είπε και η συνάδελφος από την Interact, εδώ δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με τα ιστορικά ευρωπαϊκά προγράμματα που συμμετέχουν στο εξτρατή, έχουμε και προγράμματα στα οποία συμμετέχουν οι υποψήφιες για προσχώρηση χώρες στην Ένωση. Ε, όμορας χώρας, γειτονικές μας χώρας κτλ. Και τέλος, θα ήθελα να επισημάνω επίσης τον αριθμό των εκδηλώσεων που θα γίνουν από σήμερα έως την επόμενη Κυριακή στα διάφορα προγράμματα και στα διάφορα κράτη-μέλη. Και κατά πάσα πιθανότητα σε πιο πολλές περιφέρειες από τις οποίες εσείς προέρχεστε και εκπροσωπείτε θα φιλοξενήσουν μια κάποια τέτοια εκδήλωση. Ακριβώς με σκοπό να δούμε καλύτερη προβολή στο, στην εμβέλεια αυτών των προγραμμάτων. Ο Σαν Πιέρ τώρα λοιπόν έχει το λόγο. Είστε εδώ, βλέπω, ωραία. Εκπροσωπείτε την ε, διαχειριστική αρχή του διασυνοριακού προγράμματος μεταξύ Βαλωνίας, Γαλλίας και Φλάνδρας. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα αρχικά να εκφράσω την ικανοποίησή μου που μπορώ να απευθυνθώ σε εσά ε, για να ακουστεί και η φωνή των 77 προγραμμάτων Interreg ε, στο πλαίσιο αυτής της ε, ημέρας Ευρωπαϊκή συνεργασίας. Επίση, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Μαρή Τερέ Σμιτ και το Interact. Η Βαλονία είναι μια περιοχή που είναι ανοιχτή στον κόσμο και διαμορφώνει τι δυσυνορικές σχέσει εδώ και πάνω από 20 χρόνια. Μάλιστα είναι πρωτοπόρος σε αυτόν τον τομέα, καθώς ε, από το 1988 έχει ένα πρόγραμμα με τον Νόρ καλέ», ε, το πρόγραμμα PACT και έχει αξιοποιήσει και τις δυνατότητες που προσφέρει το ΤΕΡΕΚ 1 σήμερα, επενδύει στην εφαρμογή προγραμμάτων Ευρωπαϊκής ε, Εδαφικής Συνεργασίας, τρία διασυνοριακά, ένα διεθνικό και τέσσερα διαπεριφερειακά. Εξάλλου, όπως είπε και η Πρόεδρος, η Βαλονία από το Ιντερεκ 3 και μετά είναι αρχή διαχείρισης του προγράμματος Γαλλία-Βαλονία-Φλάνδρα. Με όλη αυτή την πλούσια εμπειρία λοιπόν ήθελα να επανέλθω ε, στα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Εδαφικής ε, Συνεργασίας ε, γιατί πολύ συχνά ξεχνάμε τη στρατηγική φιλοδοξία της. Το Ιντερέκ θεωρείται συνήθως ένα χρηματοοικονομικό μέσο χωρίς στρατηγικό βάθος. Κατά τη γνώμη μου αυτό είναι λάθος γιατί ουσιαστικά ε, λέμε πώς θα διαμορφώσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα την Ευρώπη χωρίς σύνορα όπως αναφέρεται στην συνθήκη της του Μάστριχτ. Επίσης, πώς θα ε, κινήσουμε το ενδιαφέρον των ε, πολιτών για την Ευρώπη μέσω τέτοιων ε, προγραμμάτων προσέγγισης των λαών και να αναπτύξουμε την ιδέα μιας ευρωπαϊκής ηθαγένειας. Μετά, πώς θα δώσουμε μοχλούς δράσης ε, στους, ε, στις ε, παραμεθόριες περιοχές που είναι απομακρυσμένες από τους οικονομικούς πόλους και τα κέντρα λήψης αποφάσεων και βεβαίως πώς θα εκμεταλλευτούμε και θα αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες των παραμεθόριων αυτών περιοχών για να τους κάνουμε κινητήρους μοχλούς ανάπτυξης. Η συνδρομή του Interreg σε αυτούς τους πολιτικούς στόχους είναι προφανής. Το Interreg από μια απλή κοινοτική πρωτοβουλία πλέον έχει γίνει ένας από τους τρεις κύριους ε, στόχους της πολιτικής συνοχής και κατά πάσα πιθανότητα ένα από του δύο μεγάλους στόχους για την περίοδο 2014-2020. Όμως αυτή ε, η συμβολή συχνά δεν αναγνωρίζεται ε, στο ευρύ κοινό, ούτε καν πολλές φορές και στο κέντρο λήψη αποφάσεων. το, η διάδοση αυτού του προγράμματος είναι μια πρόκληση και η, η Μέρα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας μια από τις απαντήσει. Με αυτό το πνεύμα λοιπόν ε, έχουμε το δικό μας πρόγραμμα στην Ευρωπαϊκή μας Θα σας αναφέρω δύο γεγονότα, δύο εκδηλώσεις. Έχουμε μία ε, επίσκεψη στα ορυχεία που συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα Interreg ε, και πρόσφατα εντάχθηκαν και στην παγκόσμια κληρονομιά της UNESCO. Επίσης, καλούμε τους πολίτες να ανακαλύψουν το νέο κέντρο ε, διερμήνες στο στρατιωτικό ε, νεκροταφείο του Λέζεντ Χουκ ε, που βρίσκεται στο Πόπερίγκα. Θα ήθελα τώρα να σας υποβάλω κάποιες σκέψεις ό,τι αφορά τις δεσμεύσεις των σχεδίων κανονισμών αλλά και πέρα από αυτά. Οι σημερινές ρυθμίσεις ε, διαμορφώνουν και ε, επιτάσσουν μια λογική ε, οικονομική που θα βασίζεται στα αποτελέσματα. Ξέρω ότι δεν είναι κάτι καινούριο αυτό. Δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην, στην χρήση των πόρων για την επίτευξη προσθέμενης αξίας. Αυτή η αλλαγή προσέγγισης είναι ε, ευκταία όμως θα πρέπει να προσαρμοστούν και τα εργαλεία που ακολουθούμε στα προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας. Πώς όμως θα μετρήσουμε τα αποτελέσματα ε, αυτών των προγραμμάτων σε όλη την Ευρώπη αν δεν χρησιμοποιούμε τους ίδιους δείκτες και δεν συμφωνούμε επί των ορισμών. Η προσέγγιση που βασίζεται στα αποτελέσματα είναι γνωστή στον ιδιωτικό τομέα. Ε, γι' αυτό και είναι απαραίτητη η συμμετοχή του αν θέλουμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις της στρατηγικής 2020 με την ε, σύναψη εταιρικών σχέσεων δημοσίου ιδιωτικού τομέα. Για την ε, επίτευξη αυτών των στόχων λοιπόν θα πρέπει να υπάρξει και διοικητική απλούστευση. Όπως και στην Επιτροπή των Εφεριών και εμείς εκτιμούμε ότι είναι απαραίτητο να διαμορφώσουμε μια οδηγία σε ό,τι αφορά τις ε, ε, κρατικές ενισχύσεις ε, με κανόνες εντιμήνυμης ως βάση μέσω ειδικών εξαιρέσεων για τα προγράμματα αυτά θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και του ιδιωτικού φορεί ιδιαιτέρω τι μικρομεσαίες επιχειρήσει ε, στον κατάλογο των ενδεχόμενων δικαιούχων. Η συνδρομή και συμβολή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα είναι ε, ολοένα και μεγαλύτερη, καθώ θα λαμβάνει στρατηγικό ρόλο η καινοτομία στι πολιτικέ ε, συνεργασίες. Ε, αυτή, αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές, ε, αυτός ο προσανατολισμό είναι... Έχει κεντρικό χαρακτήρα στην οικονομική ανάπτυξη ζωνών συνεργασίας ε, και δεν πρέπει να ξεχνάμε το βασικό, τη βασική αποστολή του ΙΤΕΡΕΚ που είναι η διαμόρφωση μια ευρωπαϊκής ηθαγένεια. Ε, δεν πρέπει να ξεχνάμε λοιπόν αυτό το πολύ σημαντικό ρόλο του, του Ιντερεκ ε, που ανοίγει το δρόμο στην ειρήνη και στην διαπολισμητικότητα. Η συνεργασία, ε, συνίσταται βασικά στο πώς θα γνωρίσουμε ο ένας τον άλλον, πώς θα εμπιστευτούμε ο ένας τον άλλον και θα θελήσουμε να επιτύχουμε μαζί. Ε, η εξπόστο αξιολόγηση του Interreg 3 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η συνεργασία, αυτή η ήπια συνεργασία συμβάλλει και αυτή στην ε, βιώσιμη επίλυση των προβλημάτων. Εδώ έχουμε δύο λοιπόν ε, ε, οδούς, το benchmarking και την κεφαλαιοποίηση, τη δημιουργία νέων εταιρικών σχέσεων και θα πρέπει να βασιστούμε σε αυτά τα προγράμματα του Interreg. Η άλλη οδός ε, είναι το πώς θα εστιαστούμε στις ε, ε, δυνάμεις μας και θα ε, συγκεντρώσουμε τους πόρους μας. Ε, τέλος, ως εκπρόσωπος της Διαχειριστικής Αρχής θα ήθελα να κάνω, απευθύνω μια έκκληση, να τολμήσουμε περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν, να ξεπεράσουμε τους περιφερειακούς εγωισμούς για να δράσουμε προς όφελος του γενικού συμφέροντος της ε, ζώνης συνεργασίας. Σε αυτό το πλαίσιο έχει έρθει η ώρα όπου υπάρχει η πολιτική βούληση, όπου έχει οριμάσει η εταιρική σχέση, να ε, επιμηκύνουμε την ε, ε, διαδραφική συνεργασία και να, την εντάξουμε, να εντάξουμε το, το Interreg σε ένα σενάριο μετά το 2020. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ρομπέτς. Λάμπερτ Φανίστερ Ρόι. Ευχαριστώ. Από πλευρά μου και εγώ θα ήθελα να υπογραμμίσω την σημασία της συνεργασίας. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι ακριβώς τώρα με, τον νέο, με τους νέους κανονισμούς έχουμε συζητήσει επί μακρόν ε, αυτά τα σημεία, έχουμε κάνει και ακροάσεις ακριβώς ε, για αυτή την εδαφική συνεργασία στην Ευρώπη και όλα τα μέσα ε, που αφορούν αυτή τη συνεργασία έχω την εντύπωση ότι τα μηνύματα που θέλετε να στείλατε υπάρχουν ήδη στον συναδέλφων. Συμμετέχουμε σε αυτήν την εργασία λοιπόν. Όσο γίνεται περισσότερη προσοχή βεβαίω ε, δεν κάνει κακό. Ένα σημείο ήθελα να τονίσω. Δεν με ικανοποιεί ο τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται αυτά τα προγράμματα. Κάθε πρόγραμμα έχει δικό του λογότυπο. Α πάτε κάτω στην, ε- ε- στην είσοδο του Κοινοβουλίου, εκεί έχετε μια παρουσίαση του Interreg, με έξι διαφορετικά λογότυπα. Και πρέπει πραγματικά να ψάξει κάποιος για να βρει το ευρωπαϊκό λογότυπο με τα αστεράκια. Ε, ε, το Smart Specialization έχει δικό του λογότυπο, κάθε διαφορετικό πρόγραμμα έχει άλλο λογότυπο. Και αυτοί οι πολίτες, οι καημένοι, πώς ε, θα το συνδυάσουν ε, αυτή την ιδέα, ότι δηλαδή πρόκειται για πρόγραμμα συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους άλλους φορείς. Ε, έχουμε μια χιονοστιβάδα λοιπόν ε, ονομασιών και λογοτύπων. Πρέπει ε, να γίνει ένας εξορθολογισμός σε ό,τι φορά την, ε, τις ονομασίες. Εδώ και δεκαετίες συνεργαζόμαστε σε αυτό το τομέα. Βεβαίως μπορούμε να βελτιωθούμε. Πρέπει όμως να σκεφτούμε το ζήτημα της επικοινωνίας. και εδώ ίσως θα πρέπει να επιθεθούμε στους ε, συναδέλφους του Ίντερεκ, γιατί έτσι χάνεται ο κόσμος. Ε, δεν ξέρει πού να στραφεί, ουσιαστικά, ενώ ουσιαστικά πρόκειται για προγράμματα ενός, ε, μιας αποστολής Ευρωπαϊκής Συνεργασίας, Εδαφικής Συνεργασίας. με, με τα επιμέρους ε, στοιχεία των ε, περιφερειακών ε, προγραμμάτων τα κτλ. Εξορθολογισμός. Αυτό εμένα θα με ικανοποιήσει. Ευχαριστώ. Ε, ε, Ευχαριστώ πολύ. Για άλλη μια φορά θα ήθελα να πω ότι το ξεκίνημα αυτών των εκδηλώσεων γίνεται εδώ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε μια διπλάνια αίθουσα. Θα ήθελα να πω στην Μαρή Τερέ και στην Ρίκα Μάνερ που είναι η συγγήτρια και η οποία πραγματικά εργάστηκε σκληρά υπό την αιγίδα όλων αυτών που χορηγούν αυτό το γεγονός. Δεν ξέρω, Ρίκα, αν θέλεις να πεις κάτι. Σας ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά ευχαριστώ ιδιαίτερα όλους όσους οργάνωσαν ε, αυτήν την εκδήλωση. Καταρχήν την Μαριτερές, το Interact, η συνεργασία με το Interact για την προετοιμασία αυτής της έκθεσης ήταν πάρα πολύ επικοδομητική και μπορέσαμε επιτόπου να βρούμε τα στοιχεία που χρειαζόμασταν έτσι ώστε να προετοιμάσουμε τον κείμενο αυτό. Ψηφίσαμε στην Επιτροπή τον Ιούλιο και βεβαίως ε, έχουμε και την εντολή για να ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Ελπίζω αυτές οι διαπραγματεύσεις να πάνε καλά οι συνομιλίες να είναι επικοδομητικές, αλλά θεωρώ πραγματικά ότι αυτά τα προγράμματα που προωθούν και ενισχύουν αυτήν την συνεργασία είναι εξαιρετικά σημαντικές αυτήν την εποχή. Μιλάμε όλο και περισσότερο για γεφύρωμα του χάσματος και αυτού του είδους η εδαφική συνεργασία βοηθάει στην καθημερινή ζωή των πολιτών να ενισχύσουμε το συνέστημα ότι ανήκουν στην Ευρώπη. Βεβαίως πολλά πρέπει να βελτιωθούν ε, στον τρόπο που εργαζόμαστε και αυτό βεβαίως θα βοηθήσει αυτός ο κανονισμός. Χρειάζεται καλύτερη συνεργασία, αλλά κυρίως πιο απτές ε, πρωτοβουλίες, έτσι ώστε οι πολίτες να μπορούν να διαπιστώσουν ότι κάτι γίνεται στην Ευρώπη. Η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Ιούλιο ήταν σαφέστατη υπέρ αυτού του προγράμματος. Επίσης οι δημοσιονομικές δεσμεύσεις ήταν πολύ συγκεκριμένες. Υιοθετήσαμε αυτό το 7%. Η Επιτροπή είχε προτείνει 3% και πραγματικά εδώ ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους που υποστήριξαν. Γιατί όλοι κατανοήσαμε πόσο σημαντικό είναι το πρόγραμμα αυτό και βεβαίω έχουμε σήμερα μια ισχυρή βάση για τις ε, συζητήσεις μας και το Συμβούλιο. Αυτή η ημέρα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας είναι πάρα πολύ χρήσιμη για όλους. Ευχαριστώ όλους, ευχαριστώ το Interact και ελπίζω η συνεργασία αυτή να συνεχιστεί για να φτάσουμε εκεί που όλοι ευελπιστούμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους συναδέλφους. Ευχαριστώ όλους όσους εργάστηκαν σκληρά και στις 12.30 σας ζητώ όλους ε, να έρχεται έξω από την αίθουσα. Ελπίζω πραγματικά αυτή η διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ Φλάνδρας Μαλωνίας και Γαλλίας θα εμπνεύσει και πολλά άλλα προγράμματα τα οποία υπάρχουν, τα οποία έχουν ξεκινήσει ή τα οποία θα ακολουθήσουν στο ε, μέλλον. Νομίζω ότι θα πρέπει όμως να περάσουμε στις ψηφοφορίες. Ναι. Oh, να πω ότι δεν έχω την κάρτα ψηφοφορία. Το λάβουμε υπόψη, λέει πρόεδρο. Ο και ο κύριο Αγκουράκη ήθελε το λόγο, δεν σα παρατήρησα. Παρακαλώ. Θέλετε το λόγο, κύριε Αγκουράκη. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομο. Ε, ασφαλώς και τα προγράμματα στα οποία αναφερθήκαμε έχουν συμβάλει, συμβάλλουν σε θετικούς στόχους ε, και δεν είχα καμία διάθεση να αμφισβητήσω τις προσπάθειες που έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια και κυρίως ε, το τελευταίο χρονικό διάστημα. Έχω την αίσθηση όμως ότι ορισμένα πράγματα μας ξεπερνούν. Ε, υπάρχουν ορισμένες τριβές πιθανώς του χαρακτήρα της διασυνοριακής συνεργασίας όμως ε, το τεράστιο πρόβλημα και το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σήμερα στην Ευρώπη είναι, ε, και στην Ευρωπαϊκή Ένωση νομίζω είναι ο ρατσισμός και η ξενοφοβία απέναντι σε λαούς κυρίως που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παραδείγματο χάρη στην Ελλάδα άκουσα για αυτό το πρόγραμμα για τα μπουκάλια μεταξύ Ελλάδα και Ιταλία. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει κανένα που να έχει κάποιο πρόβλημα με του Ιταλού, όπω ούτε οι Ιταλοί δεν νομίζω να έχουν κανένα πρόβλημα με του Έλληνε. Όμως υπάρχει ένα θέμα που καλλιεργείται από τις άρχουσες τάξεις της Ελλάδας και της Τουρκίας μεταξύ ε- των, Ελλήνων και των Τούρκων. Ή αν θέλετε ακόμα πιο σοβαρό είναι τα προβλήματα που ξέρουμε όλοι ότι υπάρχουν σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά ε, τους μετανάστες από την άμεση γειτονιά της Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με αυτό ήθελα να πω ότι πέρα από τις προθέσεις ε, υπάρχουν ήδη πολλά πράγματα που γίνονται σε Ευρωπαϊκή Ένωση, έρασμους και διάφορες άλλες ανταλλαγές όμως πρέπει ε, πολύ περισσότερο να στρέψουμε την προσοχή μας στους μετανάστες και κυρίως στην αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων και των επιθέσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Eh, σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ας περάσουμε τώρα στις ψηφοφορίες. Να ελέγξουμε πρώτα απ' όλα τις κάρτες. Παρακαλώ βάλτε την ε, κάρτα ψηφοφορία σας. Ε, ο Μιγέλ να ξεκινήσει ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Τρεις συνάδελφοι δεν ψήφισαν, δύο. Παρακαλώ, ελέγξτε όλη την κάρτα σας. Ακόμη είναι ανοιχτή ψηφοφορία. Δύο συνάδελφοι δεν ψήφισαν. Αλλά από ό,τι βλέπω δουλεύουν ε, οι κάρτες κανονικά. Λοιπόν, πέρας ψηφοφορίες. Αν κανείς αντιμετωπίσει πρόβλημα, παρακαλώ ενημερώσει τους τεχνικούς. Ξεκινούμε με την ε, γνωμοδότηση του κυρίου Σταυρακάκη. Για την κυρία Ματσόνη το ξέρουμε, εκτός μικροφώνου όμως μιλάει η κυρία Ματσόνη. Πρόεδρος. Το κατανοώ και θα το λάβουμε υπόψη. Ξεκινάμε με Λέσλο Σούρια. συμβαστική 1, υπέρ, κατά, αποχές, Υιοθετείτε. Τροπολογία 2, υπέρ, κατά, αποχές, Υιοθετείτε. Τελική ψηφοφορία την κάνουμε ηλεκτρονικά, άρχεται ψηφοφορία. Όχι, δεν ξεκίνησε. Τώρα άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Με ευρία πλειοψηφία λοιπόν εγκρίνεται. Τώρα θα θυμάστε ότι το σημείο 13 αναβάλλεται. Πάμε στο σημείο 14 της κυρίας Κλέβα η γνωμοδότηση Ξεκινώ τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Τροπολογία 2. Χωριστή ψηφοφορία. Το πρώτο τμήμα. Ποιος είναι υπέρ. Ποιος είναι κατά. Ελέγχουμε το πρώτο τμήμα. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Υιοθετείτε έναντι 14. Λοιπόν, το δεύτερο τμήμα, Ποιο είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται, τροπολογία 3, υπέρ, κατά, υιοθετείται, τροπολογία 4, υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείται, η 5, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, τροπολογία 6, προφορική τροπολογία του εισηγητή, and local και τοπικός. Αυτή είναι η προστίκη Ψηφίζουμε υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείτε. Και ψηφίζουμε τελικά ηλεκτρονικά, άρχιτη ψηφοφορία. The vote is closed. Πέρασε. 29 υπέρ 2 κατά 3 αποχές υιοθετείτε. Τα σημεία 15 και 16 αναβάλλονται επίσης, οπότε περνάμε στην ε, ε, στο σημείο 17, έκθεση Βλάσακα. Άρχεται η ψηφοφορία. Παρακαλώ. Ναι, Πρόεδρε, για αυτή την έκθεση, πριν περάσουμε στις ψηφοφορίες, θέλω να θέσω μία ερώτηση. Υπάρχουν τροπολογίες για το άρθρο 16 Νικολάκετς. Στην Επιτροπή Ήτρε οι συντονιστές συμφώνησαν να μην υπάρξουν τροπολογίες στο άρθρο αυτό. Στον κατάλογο ψηφοφορία, λοιπόν, πολύ ορθά αναφέρεται ότι αυτό ξεπερνά τις αρμοδιότητες επιτροπές Ρέγγι. Οπότε, αν δεν είναι κανείς κατά, προτείνω οι τροπολογίες για το άρθρο αυτό να μην τεθούν στη ψηφοφορία. Και αν δεν ε, υπάρχει πλειοψηφία, να μην ψηφίσουμε κατά δύο. Δεν μιλάω για το περιεχόμενο τροπολογιών απλά γιατί δεν έχουμε την αρμοδιότητα ως Επιτροπή. Θέματα ε, ηθικής ε, στην ε, έρευνα, στη γενετική και στην εμβριολογία δεν είναι αρμοδιότητά μας. Πρόεδρος, ο κ. Βανίστερόη. Ευχαριστώ πολύ. Πράγματι δεν είναι ε, σύστημα δική μα αρμοδιότητα, ε, τα συστήματα ηθικής ε, στην έρευνα. Ίσως μπορούσαμε να το αποσύρουμε, αλλά το ΕΛΚ θα ήθελε να καταδείξει ότι στην Επιτροπή Ήτρε υποθέτω ότι θα γίνει συζήτηση, γιατί είναι πολύ σημαντικό θέμα από πλευράς ηθικής. Θα μπορούσαμε όμως να το διαγράψουμε εδώ και θα ήθελα να σημειωθεί στα πρακτικά ότι αυτό θα το επιθυμούσε η ομάδα μου. Βεβαίως θα έχουμε πολύ διαφορετική θέση σε αυτό σε σχέση με, το, με τους σοσιαλιστές δημοκράτες. Αλλά εντάξει. Ευχαριστώ. κύριος Νικολάσικ δεν είναι εδώ, αλλά με βάση τη γνώμη της Γραμματείας σχετικά με το νομικό πλαίσιο που κινούμαστε, θεωρούμε ότι αυτή η τροπολογία ξεπερνά τις αρμοδιότητες της Επιτροπής ΡΕΚΙ. Πιστεύω λοιπόν ότι έχω το δικαίωμα να ζητήσω να αποσυρθεί αυτή η τροπολογία. Και από ό,τι καταλαβαίνω υπάρχει υποστήριξη και του συντονιστή της ομάδας. Δεν ψηφίζουμε λοιπόν αυτή την τροπολογία. τώρα ξεκινάμε. Κωνσταντζα, όταν παίρνει το λόγο μετά εγώ τα χάνω, λέει ο πρόεδρο. Λοιπόν, ανθρωπολογία 23, υπέρ. Κατά, αποχές, υιοθετείτε. 24, υπέρ. Κατά, αποχές, υιοθετείτε. 25, υπέρ. Κατά, ελέγχουμε την 25. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 26 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 27 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 28 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείται. 29 υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε την 29. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 30 υπέρ. Κατά αποχές υιοθετείται 31 υπέρ. Κατά αποχές υιοθετείται 32 υπέρ. Κατά αποχές υιοθετείται. Το ελέγχουμε. Την 32 την ελέγχουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Υιοθετείται. 4 και 33. Ταυτόσημες υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. Συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές υιοθετείτε. Τροπολογία 40 υπέρ. Τροπολογία 40 επαναλαμβάνει πρώτο. κατά αποχές υιοθετείτε, 5 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. 44 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. 45 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. 47 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. 48 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. 49 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται 50 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται 51 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται 52 ψηφίζουμε γλωσσική προφορική τροπολογία είναι κανείς κατά ψηφίζουμε την 52 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται 53 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 54 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται 55 υπέρ. Κατά αποχές υιοθετείται 56 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 57 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 58 υπέρ. Κατά αποχές υιοθετείτε, 59 υπέρ. Κατά αποχές υιοθετείτε. Πάμε στα εκτιμώντας τροπολογία 6 υπέρ. Κατά αποχές υιοθετείται 7 υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείτε. 8 υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείτε. 9 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 10 υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείτε. Την 11 Τε ψηφίζουμε. Υπέρ. Κατά αποχές. Υιοθετείτε. 12. Υπέρ κατά αποχές υιοθετείται 13 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται 15 υπέρ κατά αποχές το ελέγχουμε Αφού δεν σηκώνετε το χέρι, λέει η Πρόεδρος, ελέγχουμε τη 15. Παρακαλώ, έρχεται η ψηφοφορία. Υιοθετεί τη 19, είναι τη 16. 16 ε, ε, υπέρ. Τη 16 ψηφίζουμε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε τη 16. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται, ρωτάει πρόεδρος. Απορρίπτεται. 18 υπέρ, 18 κατά. Α, μάλιστα. Συμβασμός 3 υπέρ. Κατά αποχές υιοθετείται. Τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. 18 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. Συμβασμός 4 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. 22 υπέρ κατά αποχές υιοθετείτε. Τροπολογία 3 υπέρ κατά, αποχές, υιοθετείτε. Και τελική ψηφοφορία, ηλεκτρονικά παρακαλώ, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 35 υπέρ, ε, μία ψηφοφορία κατά, συγχαρητήρια στον κύριο Βλάτσικ. Θέλετε το λόγο, να κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για τη συνεργασία σε ευχαριστούμε λοιπόν θερμά. Μια μικρή λύση για την τροπολογία 35 και 36. Να μην ψηφίσουμε δηλαδή αυτές τις τροπολογίες, συμφωνώ και εγώ, γιατί είναι εκτός αρμοδιότητας επιτροπής μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. You, colleagues, we move to point... Ευχαριστώ, συνάδελφοι. Ας προχωρήσουμε στο επόμενο το σημείο 18 για την κοινή αλληλευτική πολιτική του Γιούνου Σαματζή. Ξεκινάμε με την ε, συμβαστική 1. Υπέρ, κατά αποχές, υιοθετείται. 101. Τροπολογία 101. Υπέρ. Κατά. Να το ελέγξουμε. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 21 με 17. Τροπολογία 100. Υπέρ Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 23. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείται. Συμβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείται. 103. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείται. 104. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείται. Συμβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Να την ελέγξουμε. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Απορρίπτεται. 19 με 17. Συ... Α, συγγνώμη, τροπολογία 25. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 105. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 106 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 107 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές υιοθετείται. Συμβιβαστική 5 υπέρ. Κατά. Υιοθετείται. Συμβαστική 5 και πάλι υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. Τροπολογία 111 υπέρ, κατά αποχές υιοθετείται. Συμβαστική 6 υπέρ, κατά αποχές υιοθετείται. 115 υπέρ, κατά αποχές υιοθετείται. 116 υπέρ, κατά αποχές υιοθετείται. 117 υπέρ, κατά αποχές υιοθετείται. 118 υπέρ, κατά αποχές. Υιοθετείται 119 υπέρ, κατά να την ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. Απορρίπτεται 21 με 17. Τροπολογία 29. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 120. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Θα την ελέγξουμε την 120. Έναρξη. Πέρας. Απορρίπτεται. 19 με 17. 121 υπέρ. Κατά. Αποχές. υιοθετείται. 30 υπέρ. Κατά. Νομίζω υιοθετείται. Ας την ελέγξουμε όμως. Την 30. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας ψηφοφορίας. Υιοθετείτε. 19 με 17. Συμβιβαστική 7. Υπέρ. Κατά αποχές υιοθετείτε. 125 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 32 υπέρ. Κατά αποχές υιοθετείτε. 126 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 127 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται, 128 υπέρ, κατά αποχές υιοθετείται, 33 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 129 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 130 υπέρ, υπέρ, κατά και πάλι νομίζω απορρίπτεται, στην την ελέγξουμε την 130. Έναρξη ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορία απορρίπτεται. 131 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 132 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 133 υπέρ κατά και πάλι για την 133 υπέρ κατά αποχές υιοθετείτε, 134 υπέρ κατά αποχές υιοθετείτε, 135 υπέρ κατά νομίζω απορρίπτεται την ελέγχουμε άρχεται η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας 20-20. Άρα απορρίπτεται. 136 υπέρ. Κατά. Αποχές υιοθετείται. 137 υπέρ. Κατά αποχές υιοθετείται. 138 υπέρ. Κατά αποχές υιοθετείται. 139 υπέρ. Κατά. Να την ελέγξουμε. Έναρξη. Πέρας. Απορρίπτεται. 21 με 18. 140 υπέρ. Για την 140 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. 141 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 142 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 143 υπέρ κατά Αποχές. Απορρίπτεται. Να ελέγξουμε την 143. Έναρξη. Πέρας. 20-20. Πάλι απορρίπτεται. 144. Υπέρ. Κατά. Το μη... Νομίζω είναι το ίδιο. Ας την ελέγξουμε. Για την 144. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας ψηφοφορία. Και απορρίπτεται. 20 με 18. 146 υπέρ. Κατά αποχέ απορρίπτεται. 35 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 147 υπέρ. Κατά απόχέ ε, απορρίπτεται. 36 υπέρ. Κατά την Έναρξη. Πέρας προφορίας. Απορρίπτεται. 148 υπέρ. Κατά αποχές υιοθετείται. Συμβαστική 8 υπέρ. Κατά αποχές υιοθετείται. 151 υπέρ. Κατά αποχές απορρίτεται 152 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται 153 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται 154 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται 38 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται 39 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται 155 όχι Α, ναι. Καταπίπτει γιατί υιοθετήθηκε. 40 ε, λοιπόν υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 156 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. 41 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. 157 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. 158 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. 42 υπέρ κατά να την ελέγξουμε. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 43 υπέρ. Κατά αποχές 159 υπέρ. Κατά αποχές υιοθετείται. 165 Κατά αποχές υιοθετείται 161 υπέρ Κατά. Αποχές υιοθετείται. Όχι. Να την ελέγξουμε. Μπορεί και μια φορά να έχω κάνει λάθος. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. 21 υπέρ και 20 κατά υιοθετείται. Πού πάμε. Στην τροπολογία 50 μου λένε. Στην επόμενη σελίδα. Τροπολογία 50 για το άρθρο 34. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείται. 51. Υπέρ. 51 υπέρ. 51 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 172 υπέρ. Κατά αποχές υιοθετείται. 173 υπέρ. Κατά. Να την ελέγξουμε την 173. Έναρξη ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 174 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω το ίδιο συμβαίνει. Ας ελέγξουμε όμως για την 174. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία 22 υπέρ, 19 κατά, υιοθετείτε. 52 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 53 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται, 54 υπέρ, κατά αποχές υιοθετείται, 55 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 56 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 57 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 175 υπέρ, κατά αποχές υιοθετείται, 58 υπέρ, κατά αποχές υιοθετείται, 176 υπέρ, κατά αποχές υιοθετείται. 59 υπέρ, κατά αποχές υιοθετείται. Συμβαστική 10 υπέρ, κατά αποχές υιοθετείται. 179 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 61 υπέρ, κατά αποχές υιοθετείται. 62 υπέρ, κατά αποχές υιοθετείται εδώ ένα, υπέρ κατά υιοθετείται, εκτιμώντας δύο, υπέρ κατά αποχές ε, υιοθετείται, 63 υπέρ κατά αποχές νομίζω υιοθετείται, ας το ελέγξουμε. Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται, 25 με 15. 3 υπέρ, υιοθετείται, Συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. 65 υπέρ. 65 υπέρ. Κατά αποχές υιοθετείται. 5. Α, ελέγξουμε την 65. Έναρξη ψηφοφορίας. Α, κύριε Καρέκ, τι συμβαίνει. Πέρας ψηφοφορίας. 20 κατά 18 υπέρ. Απορρίπτεται. Τροπολογία 5 υπέρ κατά άποχες υιοθετείτε. Τροπολογία 66 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική Α, να ελέγξουμε την 66. Υιοθετείτε. 20 με 17. Συμβαστική 12 υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείτε. τερπολογιά 6 υπέρ, κατά. Δεν ξέρω για την 6, ας την ελέγξουμε. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. 21 υπέρ, 19 κατά, υιοθετείτε. 69 υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείτε. 7 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 8 υπέρ, κατά. Να την ελέγξουμε, την 8. Έναρξη ψηφοφορίας, ταεράς ψηφοφορίας, απορρίπτεται. Τροπολογία 70 υπέρ. Κατά. Αποχές υιοθετείται. Συμβιβαστική 13 υπέρ. Κατά. Αποχές υιοθετείται. 72 υπέρ. Κατά. Αποχές υιοθετείται. 73 υπέρ. Κατά. Αποχές υιοθετείται. Συμβιβαστική 14 υπέρ. Κατά. Αποχές υιοθετείται. 76 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται, 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 77 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται 78 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται όχι 78 την ελέγχουμε έναρξη πέρας ψηφορίας απορρίπτεται 12 Υπέρ. Α, συγγνώμη, 79. Υπέρ. Κατά. Δεν ξέρω για 79, να την ελέγξουμε. Έναρξη. Λήξη ψηφορίας. Απορρίπτεται. Περνάμε στη 12. Υπέρ. Τα αποχές απορρίτεται 80, 81 μάλλον, υπέρ, κατά, να την ελέγξουμε. Έναρξη ψηφοφορίας, πέρας ψηφοφορίας, υιοθετείται. 82. 82 υπέρ. Κατά. Την ελέγχουμε. Για την 82. Υιοθετείτε. 83 υπέρ. Κατά αποχές να την ελέγξουμε την 83 είναι περίεργες οι συμμαχίες σήμερα πέρας ψηφοφορίας 20-20 άρα απορρίτεται περνάμε στη 13 υπέρ κατά αποχές και πάλι ελέγχουμε. Έναρξη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Ας περάσουμε στην 85 υπέρ. Κατά. Αλέξουμε και την 85. Πέρας ψηφοφορίας. Υιοθετείτε. 14. Υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε την 14. Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται. 87. Υπέρ. κατά, αποχές, ελέγχουμε. Ακόμα και μέσα στις ομάδες ε, υπάρχουν διασπάσεις, είναι απίστευτο. Ας ελέγξουμε την 87 λοιπόν. Κλείνει, έκλεισε. Υιοθετείτε. 88 υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε την 88. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας ψηφοφορία. 21 προ 20 υιοθετείται 89 υπέρ κατά απόχέ υιοθετείται 90 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται 15 υπέρ κατά αποχές υιοθετείτε, 16 υπέρ κατά αποχές υιοθετείτε, 91 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 92 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 93 υπέρ κατά να την ελέγξουμε έναρξη Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 94 υπέρ. Κατά αποχές υιοθετείται. 95 υπέρ. Κατά αποχές υιοθετείται. 20 υπέρ. Κατά... Να την ελέγξουμε την 20. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. 21 προς 20. Υιοθετείται. 21 υπέρ κατά αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά ας την ελέγξουμε την 21. Πέρας πληροφορίας. 19 προς 19, άρα απορρίπτεται. Συμβαστική 15 υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείται για την γνωμοδότηση έναρξη ψηφοφορίας, κατά, ε, συγγνώμη, πέρας ψηφοφορίας. Και υιοθετείτε με 38 ψήφους υπέρ. Συγχαρητήρια. Ας περάσουμε στον Άντρη Κομπάτσεφ για τη θετική έκβαση τη διαδικασία έγκριση του πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου. Ξεκινάμε με την 14, τροπολογία 14. Κατά τη ονομαστική, όχι. Ψηφίζουμε λοιπόν τη 14. Εγκρίνεται. 13. Υπέρ. 13. Κατά, αποχές, εγκρίθηκε. 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 19 προφορική κατά υπέρ με την προφορική. Συγγνώμη, συγγνώμη λέει η πρόεδρος. Μου λένε ότι δεν γίνεται. Τι είπα? Α, είναι ένα, ένα τμήμα. Συγγνώμη. Συγγνώμη. Ποιος είναι υπέρ του 19. Κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα περνάμε συμβαστική 1. Υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Υπέρ. 3. Αποχές εγκρίθηκε. 4. Υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκε. 5 στην 5 αποσύρεται το δεύτερο τμήμα, άρα υπέρ του πρώτου. Κατά αποχές εγκρίνεται. 6 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 8 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 9 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 10 προφορική θα ψηφίσουμε όπως έχει τροποποιηθεί. Υπέρ 10, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα πάμε στο 11. Δύο τμήματα. Στο 11 δύο τμήματα. Αν δεν είναι κανείς κατά, ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Το δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, να ελέγξουμε το δεύτερο τμήμα, αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος, 20-20, απορρίπτεται. Και τώρα ψηφίζουμε ηλεκτρονικά, τελική ψηφοφορία, αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια. Σας ευχαριστώ πολύ. Point 23, which was this afternoon, is the, is the point of order. Of what? Colleagues, Συμφωνήσαμε με τους Κιώδης και με τον εισηγητή, ιδιαίτερα με τους Κιώδης, θα σας πω γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό, ότι τώρα θα περάσουμε στο 23. Μπορείτε να παραμείνετε, γιατί είναι δύσκολο το θέμα. Ίσως ακούσατε ότι ο κύριος Ομάρ Τζίχου που ήταν εισηγητής για την κοινή οργάνωση των αγορών γεωργικών προϊόντων εγκαταλείπει την προσπάθεια να μας παρουσιάσει εδώ ένα σχέδιο γνωμοδότησης. Βρισκόμαστε λοιπόν στην εξής κατάσταση. Αν δεν υπάρχουν τροπολογίες από τους κοιόδης, τότε πρέπει να στείλω μια επιστολή στην Επιτροπή Γεωργίας λέγοντας ότι δεν γνωμοδοτούμε. Αν όμως υπάρχουν τροπολογίες οι οποίες έχουν υποβληθεί από τους κοιόδης, τότε θα στείλουμε την γνωμοδότησή μας παρόλα αυτά. Απλώς σας το λέω για να καταλάβετε ποια είναι η κατάσταση. Κύριο Μαρζή, μπορείτε να μας εξηγήσετε πώς έχει η κατάσταση. Μπορείτε να αιτιολογήσετε τη θέση σας. Έχετε το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω τους συναδέλφους καταρχήν όσον αφορά την ψηφοφορία. Είδατε ότι ήταν πάρα πάρα πολύ κοντά το αποτέλεσμα. Τελικά όμως καταφέραμε μέσω των συμβιβασμών να επιτρέψουμε να περάσει το κείμενο για την κοινή αλληλευτική πολιτική. Τώρα, όσον αφορά το άλλο θέμα, την κοινή οργάνωση των αγορών γεωργικών προϊόντων. Εδώ πρόκειται για μια γνωμοδότηση. Επί της ουσίας αρμόδια είναι η Επιτροπή Γεωργίας. Πρόκειται για την κοινή οργάνωση των αγορών ε, τόσο της ζάχαρης, ε, το γάλατος αλλά και του ίνου. Καταλαβαίνω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για ε, τη γεωργία το θέμα αυτό. Έχω υποβάλει πάρα πολλές τροπολογίες στην Επιτροπή Γεωργίας αλλά επειδή πρόκειται να γνωμοδοτήσουμε εκ μέρους της ε, Περιφερειακής Επιτροπής, έχω πρόβλημα όσον αφορά την σχέση που έχουμε. Αλλιώς βεβαίως θα έπρεπε να προετοιμάσω ένα θεωρητικό κείμενο, κάτι το οποίο δεν είναι δική μου αρμοδιότητα. Ε, επειδή λοιπόν πρόκειται για ένα καθαρά συγκεκριμένο γεωργικό θέμα, θα ήθελα να σας ζητήσω να υποβάλλετε τροπολογίες. Εκτός εάν κάποιος εδώ θεωρεί ότι υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ του δικού μας αντικειμένου και του θέματος αυτού. Πρόεδρος, θα δώσω το λόγο στους Κιώδης. Α, η Κωνσταντζα. Ναι, είναι λίγο περίεργη αυτή η κατάσταση. Κανονικά οι σκιώδεις αποφασίζουν αν ναι ή όχι θα κάνουμε έκθεση ή θα κάνουμε γνωμοδότηση. Και εγώ ξέρω ότι εδώ θα μπορούσε να είχε πάρει άλλη απόφαση η Επιτροπή και θα είχαμε συμφωνήσει αν το θέμα αυτό είχε συζητηθεί στους σκιώδες μεταξύ των ε, σκιωδών εισηγητών. Τι να σας πω, δεν καταλαβαίνω. Μπορούμε να στείλουμε μία επιστολή και ενδεχομένως ε, οι συνάδελφοι αν θέλουν να στείλουν τις τροπολογίες τους κατευθείαν στην Επιτροπή Γεωργίας. Αυτή είναι η άποψη των σοσιαλιστών από ό,τι καταλαβαίνω. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να ακούσουμε τους σκιώδεις. Αν οι σκιώδεις θέλουν να συνεχίσουν, θα υποβληθούν τροπολογίες και μπορούμε από νομικής απόψεως να το κάνουμε εξ ονόματος της Επιτροπής. Η δεύτερη άποψη είναι αυτή που προτείνει η κυρία Κρέλ. Δεν ξέρω αν κάποιος άλλος θέλει να πάρει το λόγο. Σαμ Κέλλη. Ναι, καταλαβαίνω αυτό που λέει ο κύριος Σομάζη. Είναι παράδοξο και πολύ καθυστερημένο το θέμα και όπως ε, το αντιμετωπίζουμε. Βεβαίως είναι κάτι το οποίο μπορεί να το ξαναντιμετωπίσουμε. Είναι σημαντικό το θέμα πάντως της έκθεσης αυτής και σαφώς και επηρεάζει όλα τα κράτη-μέλη. Έχει συνέπειες. Γι' αυτό και είναι σημαντικό τουλάχιστον να υποβάλουμε κάποιες τροπολογίες. Έτσι τουλάχιστον δείχνουμε ότι δραστηριοποιούμεθα για το θέμα αυτό και μπορούμε, εν πάση περιπτώσει, να επηρεάσουμε το θέμα αυτό. Ας θέσουμε λοιπόν μία προθεσμία για την υποβολή των τροπολογιών. Αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να κάνουμε. Ευχαριστώ. Ο Λούις. Ευχαριστώ Πρόεδρε ήθελα να πω ότι πράγματι αυτό το θέμα είναι πυρηνική σημασία, αν μάλλον είναι στον πυρήνα της ε, ουσίας της κοινή αγροτικής πολιτικής. Είναι από του μηχανισμού βάσει του οποίου οι αγρότε και η κοινή αγροτική πολιτική ε, θα επιτρέψει να υπάρξουν εισοδήματα στο μέλλον και ταυτόχρονα όμως χαρακτηρίζεται από ένα σαφή πολιτικό προσανατολισμό. Είναι σίγουρο λοιπόν ότι ο αντίκτυπος θα είναι μεγάλο σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Για αυτό το λόγο η λύση που εξευρέθηκε, δηλαδή να παραμείνουν ανοιχτές ε, οι πόρτες για κάποιους τροπολογίες που αφορούν τις περιφερειές μας και αυτή αν θέλετε η διαφυγική προσέγγιση ε, στην οργάνωση της κοινή οργάνωσης αγοράς ώστε να έχουμε καλύτερη προστασία κάποιων έθραυστων ζωνών θεωρούμε ότι είναι κάτι που πρέπει να παραμείνει να μην είναι ανοιχτό αυτό το παράθυρο και θεωρώ ότι είναι μία λύση και υπερασπίστηκε και ο συντονιστής της σοδεστικής ομάδας, ο Ακραίο, έκανε, ήταν μια πολύ καλή επιλογή. Θεωρούμε ότι και κάποιες άλλες προτάσεις προς αυτήν την κατεύθυνση ακριβώς πρέπει να υποστηριχθούν. Ευχαριστώ. Καταλαβαίνω ότι οι υπόλοιποι συντονιστές δεν είναι εδώ. Δεν είναι εδώ αυτοί που ήταν χτες εδώ. Εν πάση περιπτώσει, καταλαβαίνω ότι οι εισηγητές θέλουν να συνεχίσουν. Αυτό καταλαβαίνω. Θέλετε να υποβληθούν τροπολογίες. Ας θέσουμε λοιπόν κάποια ημερομηνία και να συνεχίσουμε. Στέλνοντας μία επιστολή στην Επιτροπή Γεωργίας. Με αυτόν τον τρόπο θα στείλουμε τις τροπολογίες που θα υποβάλουν και οι σκιώδεις, αλλά και όλοι όσοι επιθυμούν να το κάνουν. Θέλετε να πάρετε το λόγο επί της ουσίας σήμερα. Όχι. Ωραία. Διευκολύνουμε την διαδικασία. Αντί να στείλει ο καθένας ε, μόνος του τις ε, τροπολογίες ουσιαστικά τις συγκεντρώνουμε και θα τις στείλουμε σαν Περιφερειακή Επιτροπή. Πρέπει να ψηφίσουμε τον Οκτώβριο, άρα η υποβολή των τροπολογιών πρέπει να γίνει πολύ γρήγορα. 20. Σε δύο μέρες δηλαδή. 20 Σεπτεμβρίου το μεσημέρι. 12. προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών. Τελειώσαμε και με το θέμα αυτό. Δυστυχώ. επειδή ήμασταν πάρα πολύ γρήγοροι στι τροπολογίες, θα πρέπει να περιμένουμε στις 11 που θα έρθει ο Επίτροπος. Έχουμε λοιπόν χρόνο στη διάθεσή μας. Μπορούμε να περιμένουμε. Δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω το χρόνο αυτό για κάτι άλλο. Έχω κάποιες ανακοινώσεις τις οποίες δεν έκανα χτες, διότι ο Επίτροπος ε, βιαζόταν πάρα πολύ. Μπορώ λοιπόν να σας ενημερώσω όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις. Θυμάστε φαντάζομαι ότι τον Ιούλιο δώσαμε εντολή για διαπραγματεύσεις. Αφήσαμε παρόλα αυτά κάποια θέματα, ιδιαίτερα αυτά που αφορούν τον δημοσιονομικό κανονισμό θα ήθελα να σας ενημερώσω λοιπόν ότι οι υπόλοιπε εντολές που αφορούν αυτόν τον κανονισμό, καθότι και τις ιατρολογικές σκέψεις, οι εντολές αυτές θα δοθούν τον Νοέμβριο. Θα ήθελα επίσης να σας ενημερώσω ότι θα ξεκινήσει η τριμερής συζήτηση με την Επιτροπή και με το Συμβούλιο. Έχουμε συμφωνήσει όσον αφορά τη μέθοδο εργασίας, τους έχουμε ενημερώσει για το πώς θα οργανώσουμε τις ομάδες διαπραγμάτευσης. Συμφωνήσαμε ότι η διαπραγμάτευση θα γίνει βάση του εγγράφου περιλαμβάνει αυτές τις τέσσερις ε, στήλες με τις συμβιβαστικές ε, προτάσεις, ότι οι διαπραγματεύσεις θα γίνουν ε, βάσει κάποιων πακέτων, blocks. Από ό,τι φαίνεται, το πρώτο πακέτο, μπλοκ που θα διαπραγματευτούμε αρχές Οκτωβρίου, θα αφορά την στρατηγική προσέγγιση και κατόπιν θα ακολουθήσει μια θεματική συζήτηση, προσέγγιση. Αυτό όσον αφορά τη μορφή των διαπραγματεύσεων. Επίσης θα ήθελα να σας πω ότι όλα αυτά τα μπλοκ διαπραγμάτευση, τα θέματα, όλα αυτά είναι ενδεικτικά. Καθότι ξέρετε ότι μπορεί να παρεκκλίνουμε από αυτή τη μέθοδο εργασία. Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά είναι ενδεικτικά, αλλά από ό,τι φαίνεται όλοι επιθυμούν να επιταχύνουμε τις διαδικασίες και τα τρία θεσμικά όργανα. Θα ήθελα επίσης να σας υπενθυμίσω ότι η απόφαση της συνδιάσκεψης των Προέδρων είναι ότι δεν μπορούμε ατομικά σαν επιτροπή ενώ να ζητήσουμε να πάει ένα θέμα στην Ολομέλεια, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε την απόφαση των Προέδρων. Όταν δηλαδή το θέμα είναι όριμο για να πάει στην Ολομέλεια, καθότι υπάρχει σχέση ε, άμεση μεταξύ των διαπραγματεύσεων για το δημοσιονομικό πλαίσιο και για τα νομοθετικά θέματα. Καταλαβαίνετε λοιπόν δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε μια συμφωνία από τη στιγμή που άλλες συμφωνίες εκρεμούν, δεν έχουν προχωρήσει αρκετά κτλ. κτλ. Ελπίζω ότι αυτό δεν θα μας επιβραδύνει. Αυτά πάντως είναι αυτά που αποφάσισαν οι πρόεδροι. Επίσης συμφωνήσαμε ότι όταν δεν υπάρχει πρόεδρος για να προεδρεύσει αυτές τις διαπραγματεύσεις, τότε οι εισηγητές είναι αυτοί οι οποίοι προεδρεύουν των διαπραγματεύσεων. Να σας πενθυμίσω πίσω τον Ιούλιο αποφασίσαμε οι εισηγητές έρχονται στις επιτροπές, ενημερώνουν σε τακτικά χρονικά διαστήματα. Η ενημέρωση δηλαδή είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνεται οργανωμένα και για να υπάρχει καλύτερος συντονισμός μεταξύ των διαφορετικών διαπραγματεύσεων μεταξύ των διαφορετικών κανονισμών για να διασφαλίσουμε δηλαδή έναν πιο αποτελεσματικό συντονισμό και συνοχή μεταξύ των ε, διαφόρων θεμάτων, συμφωνήσαμε χτες ότι οι συγητές θα μπορούν να παρίστανται και σε διαπραγματεύσεις άλλων που αφορούν άλλους κανονισμούς. Κάτι το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο ή να είναι απαραίτητο. Αυτό λοιπόν και κάτι άλλο που θα ήθελα να σας πω. Όσον αφορά το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, οι διαπραγματεύσεις γίνονται ξεχωριστά. Σήμερα όμως η Κυπριακή Προεδρία θα κάνει την παρουσίασή της χωρίς όμως να παρουσιαστούν νούμερα. Για πρώτη φορά το Νοέμβριο θα παρουσιαστούν τα ε, νούμερα 22-23 Νοεμβρίου στη συνάντηση κορυφής για το δημοσιονομικό, πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Προτείνονται κάποιες περικοπές στο προϋπολογισμό, όπως ξέρετε, και για την πολιτική συνοχής. Εγώ ενημερώνω όλους τους συναδέλφους και ελπίζω να κάνετε και εσείς το ίδιο ότι η πολιτική συνοχής ήδη έχει υποστεί δύο μεγάλα κύματα περικοπών. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή κάτω από τα ποσά που είχαν αρχικά αποφασιστεί. 5 δις επιπλέον περικοπές και αν ακολουθήσει και άλλη περικοπή, καταλαβαίνετε ότι οι πολιτικοί συνοχής και αυτά τα λέω σε σχέση με τα σημερινά ποσά. Η θέση του Κοινοβουλίου, και γι' αυτό σας τα λέω αυτά, πριν από ένα χρόνο, βάσει της έκθεσης ΣΟΥΡ, η απόφαση του Κοινοβουλίου ήταν να παραμείνουμε στα επίπεδα. Ήδη λοιπόν έχουν ακολουθήσει δύο σημαντικές περικοπές παρόλοι που η άποψη του Κοινοβουλίου ήταν διαφορετική. Τα πράγματα λοιπόν δεν είναι απλά και θα πρέπει όλοι να χρησιμοποιήσουμε τις ευκαιρίες που έχουμε έτσι ώστε να ενημερώσουμε. Καθότι έχουμε και τη δήλωση του Συμβουλίου ότι η πολιτική συνοχή είναι μια πολιτική ανάπτυξης και ιδιαίτερα σήμερα στην ε, περίοδο που βρισκόμαστε είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Αυτές λοιπόν οι περικοπές δεν ανταποκρίνονται σε αυτήν την ε, γενική δήλωση. Η Προεδρία της Κύπρου τον Αύγουστο έκανε κάποιες δηλώσεις. Σας ζητώ, εάν δεν το έχετε κάνει ήδη, να διαβάσετε αυτές τις δηλώσεις προτείνοντας να γίνει ένας σαφής διαχωρισμός μεταξύ των νομοθετικών ε, προτάσεων και όσον αφορά την συναπόφαση να μην ε, υπάρξει καμία ανάμειξη με τις αποφάσεις που λαμβάνονται στα πλαίσια του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου. Αυτά όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις που αφορούν το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Στην πράξη θα πρέπει οπωσδήποτε να περιμένουμε και τους αριθμούς. Κάτι το οποίο μας υποχρεώνει να περιμένουμε αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να αντιδράσουμε αν δεν έχουμε συγκεκριμένου αριθμού. Δεν ξέρω αν θέλετε να πάρετε το λόγο. Ναι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μια ερώτηση. Ίσως δεν κατάλαβα καλά τι είπατε. Μπορείτε να με βοηθήσετε να κατανοήσω καλύτερα. Ποια θα είναι η διαδικασία για τον τρομερή διάλογο. Αν κατάλαβα καλά, έχουμε τη διαπραγματευτική ομάδα Αλλά την επόμενη Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει διαπραγμάτευση για το Γενικό Κανονισμό, τον εισηγητή του Γενικού Κανονισμού. Οι άλλοι εισηγητές θα προσκληθούν, αν είναι αναγκαίο, για τη διαπραγμάτευση του Γενικού Κανονισμού. Άρα, τι περιμένουμε να συζητηθούν οι άλλοι κανονισμοί σε άλλο τριμερή διάλογο ή θα γίνουν παράλληλα οι συζητήσεις. Ρωτώ. Έχουμε δηλαδή μια πρώτη ζήτηση τώρα για αυτόν τον κανονισμό και μετά θα ακολουθήσουν άλλε προσκλήσει για του άλλου ηγητέ. Ή θα γίνουν παράλληλε πραγματεύσει. παρακαλούμε, για να προετοιμάσουμε την ατζέντα μα, να μην χαθούμε. Ευχαριστώ πολύ, λέει Πρόεδρο. Τώρα όλα αποφασίζονται. Η προσέγγιση γενικά είναι ότι επειδή ξεκίνησαν οι συζητήσει για, το γενικό, ε, για το γενικό κανονισμό, συγγνώμη, καθώ εκεί λαμβάνονται γενικότερες αποφάσεις που θα επηρεάσουν και άλλου τομεακού κανονισμού, Γι' αυτό το κάνουμε έτσι, αλλά δεν έχουμε την πολυτέλεια να κλείσουμε πρώτα απ' όλα το γενικό κανονισμό για να περάσουμε στους υπόλοιπους. Προσπαθούμε λοιπόν να βρούμε ποιος είναι ο καλύτερος δυνατός συνδυασμός ώστε να γίνονται ε, με τον καλύτερο τρόπο και οι δύο διαπραγματεύσεις και για, τον, για τους και για το γενικό ε, κανονισμό. Όταν θα μπούμε τώρα στην ουσία των διαπραγματεύσεων, που αν δεν κάνω λάθος ξεκινά στις 2 Οκτωβρίου για το γενικό κανονισμό, τότε θα ξέρουμε καλύτερα τα πλέον σημαντικά ζητήματα ε, για τομεακά ζητήματα θα προκύπτουν στη συζήτηση. Οπότε θα κάνουμε ένα γενικό σχεδιασμό και να δούμε πώς μπορούμε να έχουμε τις συνδέσεις και τις ταυτίσεις για τα ζητήματα και έπειτα πριν από κάθε συνάντηση με αντικείμενο το γενικό κανονισμό θα βλέπουμε τα επιμέρους θέματα ώστε να δούμε κατά πόσον και οι συγκητές για τομεακά ζητήματα είναι σημαντικό να είναι παρόντες. Και το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι ότι Περιμένουμε τώρα τις προτάσεις σας. Η γραμματεία και εμείς θα κάνουμε την πρώτη συνάντηση για να διαθρώσουμε τις διαπραγματευτικές ομάδες. Ελπίζω ως αρχές Οκτωβρίου να έχουν κλείσει αυτά, οπότε αυτή τη στιγμή λιγάκι υπομονή. Και από εκεί πέρα θα δούμε ακριβώς πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα το χρόνο και θα προσκαλέσουμε αναλόγως τους εισηγητές των τομιακών κανονισμών. Θα δούμε λοιπόν πώς μπορούμε να ε, οδηγήσουμε όσο είναι πιο ομαλά τα πράγματα. Αλλά δεν μπορώ να σας πω εγώ ότι στις 28 Οκτωβρίου θα δοθούν οι προσκλήσεις και για το Περιφερειακό Ταμείο. Δεν μπορώ να σας πω αυτό, αλλά υπάρχει μια ισχυρή βούληση και στο Συμβούλιο και στην Κομισιόν, αλλά ιδίως στο Κοινοβούλιο, να έχουμε έναν καλό συντονισμό το κατά πόσο αρκεί αυτό να γίνει μέσω ομάδα εργασία θα το δούμε. Εγώ πιστεύω ότι είμαστε ρεαλιστέ και να προβλέψουμε τη συμμετοχή των α, εισηγητών για τους τομεακούς κανονισμούς όποτε είναι αναγκαίο και στις διαπραγματεύσεις για τον γενικό κανονισμό που θα πρέπει όχι μόνο για να ακούσουν τις συζητήσεις αλλά και για να πούν την απόψή τους. Χρειαζόμαστε όμως λίγο χρόνο παραπάνω. Όμως θέλω να σας καθησυχάσω ότι τα πράγματα τώρα είναι πιο ανοιχτά και υπάρχει ε, καλύτερη συνεννόηση και άλληλο ε, κατανόηση σχετικά με το πώς μπορούν να κυλήσουν καλύτερα οι διαπραγματεύσεις. Ο Λαμπέρ. Ευχαριστώ πολύ για όλες τις πληροφορίες. Ένα μικρό σημείο μόνο. Ε, αυτή η συζήτηση για τα στοιχεία. Έχουμε την έκθεση, τη θέση μας, την έκθεση και όλα αυτά. Θα υπάρχουν όμως ε, γρήγορες εξελίξεις στη συνέχεια. Ε, ότι δηλαδή στα αρχές Νοέμβρη το Συμβούλιο θα μας δώσει στοιχεία. Ποιος θα είναι ο ρόλος μας τότε, γιατί θα υπάρχει μια ενδιάμεση έκθεση. Και ποια είναι η θέση της Επιτροπής μας τότε. Στι αρχές του Νοεμβρίου θα έχουμε τα στοιχεία, τέλη Νοεμβρίου το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο θα ε, ε, πάρει θέση στην Ολομέλεια. Όμως πώς θα προετοιμάζουμε όλα αυτά, μπορούμε να επιταχύνουμε, έχουμε χρόνο να ε, συντάξουμε γνωμοδότηση ε, στην Επιτροπή ε, Προπολογισμού. Εμεί είμαστε διατεθειμένοι να συμβάλλουμε, ιδίω αν υπάρχουν τα στοιχεία. Και αμέσως μετά όλοι θα αρχίσουν να μιλάνε για τα στοιχεία, για τα θεωρητικά στοιχεία. Ενώ προ το παρόν δεν έχουμε την δυνατότητα να τι, συμβαίνει. Πρώτα απ' όλα, τα μοναδικά αριθμητικά στοιχεία που υπάρχουν στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου είναι αυτά της Επιτροπής ΣΟΥΡ. Και δεν ε, υπάρχει πρόταση να αλλάξουν σε αυτό το στάδιο. Δεύτερον, η Επιτροπή Προπολογισμού προετοιμάζει την ενδιάμεση έκθεση ήταν διάφορες ημερομηνίες, νομίζω κάποια στιγμή στον Οκτώβριο θα γίνει αυτό και σε αυτή την... Ε, η δομή αυτής της ενδιάμεσης έκθεσης είναι άγνωστη, αλλά πρέπει να έχουμε κατά νου ότι το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο είναι κανονισμός του Συμβουλίου που θα μας σταλεί. Ε, ο κανονισμός του Συμβουλίου είναι κάτι πολύ περιορισμένο γιατί μας δίνει απλώς επικεφαλίδες, ε, δεν μας δίνει περαιτέρω λεπτομέρειες. Και από ό,τι κατάλαβα η ενδιάμεση έκθεση που προετοιμάζει η Επιτροπή Προπολογισμού, την ίδια φιλοσοφία πρέπει να σέβεται. Γιατί αν βάλουμε σε αυτή την ενδιάμεση έκθεση όλα αυτά τα στοιχεία και να εμβαθύνουμε ε, στον προπολογισμό, τότε συμφωνούμε ότι ο κανονισμός ε, του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου πρέπει να έχει αυτά τα στοιχεία. Επομένω, εγώ αναμένω ότι η ενδιάμεση έκθεση ουσιαστικά θα αντικατοπτρίζει τις ε, θέσεις μας ε, για το τι, σε τι συνίσταται αυτό το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο του Συμβουλίου και δεν πρέπει να ε, συγχαίεται με την νομοθετική πρόταση. Δεν πρέπει λοιπόν να το βάλουμε στην ενδιάμεση έκθεση εφόσον ανήκει στην νομοθεσία. Όμως ίσως κάποιο παράρτημα να σημαίνει αυτό, γι' αυτό πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί ε, σε όλα τα βήματα και όσοι από εσά συμμετέχετε στην Επιτροπή Προπολογισμού και ενδεχομένω να παρίσταστε και εκεί, ε, να ε, προωθήσετε και τα συμφέροντα της Επιτροπής της Περιφερειακής. Να φροντίσετε τους ώστε να συζητηθούν τα, θέματα που μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερως. στην ομάδα επαφών στην οποία συμμετείχαμε τον πρόεδρο και ήμασταν όλοι οι διαπραγματευτέ. Ε, είμαστε σε αυτό το στάδιο που δεν υπάρχουν νέε πληροφορίε αυτή τη στιγμή, αλλά καθίσταται σαφέ από ε, τι ε, ομιλίε και δηλώσεις του Προέδρου του Κοινοβουλίου ότι πρώτα πρέπει να ψηφίσουμε την γνωμοδότηση για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και μόνο τότε θα μπορέσουμε να βάλουμε τα αριθμητικά στοιχεία στο νομοθετικό πλαίσιο. Πρέπει λοιπόν να περιμένουμε για την... Ε, Περιμένουμε να φτάσουμε λοιπόν σε αυτό το στάδιο των διαπραγματεύσεων για το πολιτές δημοσιονομικό που να μπορούμε να βάλουμε για τα στοιχεία. Γιατί δεν μπορούμε να ε, ε αποκλείσουμε και το γεγονός, ε, το εδεχόμενο του βέτο. Ε, μπορεί το Κοινοβούλιο να μην ικανοποιηθεί από την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων. Να ελπίσουμε ότι δεν θα συμβεί αυτό. Κάτι ακόμα, οι συνάδελφοι που θεωρούν ότι αρκεί να μπλοκάρουμε τα στοιχεία και θα μπλοκάρουμε το πολιτές πλαίσιο γιατί ο προπολογισμός του 2013 θα ε, αναπαραχθεί στο μέλλον. Αν όμως δεν έχουμε νομική βάση να ε, ξεκινήσουμε τα καινούργια προγράμματα πολιτικής, δεν ε, έχει σημασία αν θα υπάρχουν χρήματα ή όχι. Και πάλι Ακόμα οι νομικέ υπηρεσίε ε, εργάζονται σκληρά για να δουν αν μπορούμε να περπαιδίσουμε αυτό το πρόβλημα της ε, έλλειψης νομικής βάσης για την εφαρμογή των ε, πολιτικών, αν υπάρχει ο προπολογισμό ο προσωρινός για το 2013. Στα επίπεδα του 2013, ενώ δεν υπάρχει συμφωνία για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Μένει ανοιχτό όμω αυτό το θέμα. δεν μπορούμε να πούμε ότι αποδεχόμεθα τα επίπεδα προπολογισμού του 2013 και προχωράμε, γιατί δεν έχουμε νομική βάση. Περιμένουμε τον Επίτροπο τώρα. Ελπίζουμε να βρίσκεται καθοδόν. Ας κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Αγαπητοί συνάδελφοι, να ξεκινήσουμε την ε, συνάντησή μας με τον ε, Επίτροπο Γιώχανες Χάν. Έχουμε μία μισή ώρα στη διάθεσή μας για αυτή τη συζήτηση, για ερωτήσεις, παρατηρήσεις. Θα ήθελα όμως να σας παρακαλέσω να είστε όσο δυνατόν πιο σύντομοι στις παρεμβάσεις σας. Δεν ξέρω τι θέλει να μας πει ο Επίτροπος. Ελπίζω να είναι σημαντικά και ενδιαφέροντα τα όσα έχει να μας πει και να συνδέονται ε, με το τρέχον στάδιο των εργασιών μας ε, για το μέλλον της πολιτικής συνοχής. Ε, Επίτροπε, έχετε τον λόγο και ελπίζω τώρα να είστε σε θέση και να έχετε το σθένος να αντιπαλέψετε όλους τους άλλους στην Επιτροπή που έχουν αντιθέσει με εσάς. Ευχαριστώ, Νανοδά. Ευχαριστώ και εγώ και σας καλωσορίζω όλους. Θα ήθελα να προσπαθήσω και εγώ να μιλήσω σύντομα. Ξέρω ότι εχθές μιλήσατε με τον Αντιπρόεδρο τον Επίτροπο Κάλλας. Εγώ θα μιλήσω για την διευκόλυνση ε, αυτή που προβλέπουμε στην ε, Ευρώπη. Ξέρω ότι υπάρχουν ήδη κάποια στοιχεία τα οποία τα γνωρίζετε. Είμαι στη διάθεσή σας βεβαίως και για ε, ερωτήσεις. Όλοι ξέρουν βεβαίως ότι υπάρχει αυτό το ποσό, τα 10 δις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει εδώ όμως μια σαφής διάκριση μεταξύ των ε, προθέσεων, των στόχων και της υλοποίησης. Και βεβαίως το non-paper της Επιτροπής και όλες οι απτές, αν θέλετε, στην πράξη συνέπειες, σαφώς και θα πρέπει να μας απασχολήσουν περισσότερο. Οι αρμόδιοι φορείς εδώ θα πρέπει να παίξουν τον ρόλο τους. Εμείς ε, έχουμε έναν πολύ συγκεκριμένο ρόλο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ε, υπάρχει το νομοθετικό κομμάτι και υπάρχει το πάρα πολύ σημαντικό της υλοποίησης και βεβαίως ε, των διαθέσιμων πόρων, μέσων και προσωπικού. Θα πρέπει εδώ βεβαίως το σύστημα να γίνει σαφές και να μην βασιστούμε στην αρχή του όποιος προλάβει ε, θα πάρει την χρηματοδότηση. Θα πρέπει να υπάρχει μια σαφής ρύθμιση, κανονισμοί για τις διαδικασίες αυτές. Μιλάμε για ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, δίκτυα ενέργειας, δίκτυα μεταφορών, ICT και φυσικά αυτό που είναι εδώ σημαντικό είναι ότι έχουμε πάρα πολλές δυνατότητες συμβιβασμού. Και αυτό είναι αυτό που θα πρέπει να ε, προσπαθήσουμε όλοι, να βρούμε τρόπους να καλύψουμε τις περισσότερες ανάγκες των πολιτών της Ευρώπης. Ξέρω ότι έχουν ήδη ακουστεί σχόλια για τις δικές σας αποφάσεις. Επιτρέψτε μου και εγώ να πω ότι πραγματικά η Επιτροπή Ρέγγι οι ε, πρόεδρος, οι εισηγητές, όλοι όσοι συνεργάστηκαν, θα πρέπει εδώ να τους ευχαριστήσω. Οι συζητήσεις ξεκίνησαν σε μια επικοδομητική βάση και όσον αφορά τις απόψεις ε, της Επιτροπής ε, Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να μπούμε σε κάποιες αποσαφηνήσεις και επί του περιεχομένου και νομίζω δεν θα ξαφνιαστείτε αν ακούσετε ότι και εγώ αλλά και οι υπηρεσίες μου δεν θα ακολουθήσω 100% όλες σας τις απόψεις και αποφάσεις. Νομίζω ότι αυτό θα σας ξάφνιαζε εξάλλου αν συνέβαινε. Αλλά πρέπει να σας πω ότι σε μεγάλο βαθμό υποστηρίζω και συμφωνώ ε, με αυτά τα οποία πρεσβεύεται. Πιστεύω επίσης ότι μπορούμε να βρούμε μια κοινή ε, κατεύθυνση, έναν κοινό προσανατολισμό για το πού θέλουμε να οδηγήσουμε αυτήν την περιφερειακή πολιτική. Ένας κώδικας συμπεριφοράς, μια δεοντολογία η οποία θα μας οδηγήσει σε καλύτερη συνεργασία και αυτό σε πολλά επίπεδα είναι πάρα πολύ σημαντικές λοιπόν εδώ οι θέσεις ε, και οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά την περαιτέρω διαπραγμάτευση που θα έχουμε με το Συμβούλιο, που θα έχετε με το Συμβούλιο. Ε, υπάρχουν σαφείς προϋποθέσεις που έχουν ε, βεβαίως ε, τεθεί και στον τομέα του κοινού στρατηγικού πλαισίου η Επιτροπή τις τελευταίες, ε, τις τελευταίες αυτές ημέρες έχει υποβάλει μια συμβαστική ε, πρόταση με σκοπό να βρεθούν ε, υλοποιήσιμες λύσεις και πιστεύω ότι και το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να εξετάσει εδώ όλες τις δυνατότητες να δικτυωθεί το κείμενο αυτό και σε σχέση με τους υπάρχοντες κανονισμούς, αλλά βεβαίως εδώ θα αναφερθώ και στην κατεξουσιοδότηση πράξη, γιατί πιστεύω ότι εδώ πρέπει οπωσδήποτε να βρούμε μια λύση και ε, σχετικά γρήγορα. Τώρα, σε ποια σημεία διαφωνώ ή έχω διαφορετική άποψη. Αυτά πρέπει να τα συζητήσουμε βεβαίως, αλλά υπογραμμίζω, για να μην έχετε λανθασμένη εντύπωση, Σκοπός μου δεν είναι να επιμείνω στα σημεία αυτά, γιατί στα πιο πολλά μπορώ να συμφωνήσω. Ένα σημείο το οποίο δεν μπορεί να με βρει 100% σύμφωνο είναι το θέμα της θεματικής συγκέντρωσης. Οι διαφορετικές απόψεις, ε, οι διαφορετικές ε, αποφάσεις που βασίζονται στην θέση του Κοινοβουλίου ε, δίνουν την εντύπωση ότι κατά κάποιο τρόπο συγχέεται ή αποδυναμώνεται αυτό το θέμα της ε, θεματικής συγκέντρωσης. Και νομίζω ότι εδώ πρέπει πραγματικά να ακούσετε την άποψη της Επιτροπής, έχουμε δείξει αρκετή ευελιξία θα έλεγα έτσι ώστε να ενσωματωθούν θέματα όπως ε, ICT ε, και βεβαίως έχουμε θέσει σαφέστατα και εμείς κάποιες θεματικές προτεραιότητες, κεντρικά σημεία όπως ε, μεταφορές σε αστικές περιοχές, απόδοση στον τομέα της ενέργειας, μέτρα συγκεκριμένα τα οποία βεβαίως χρειάζονται περισσότερη συζήτηση. Αλλά αν προσθέσουμε και άλλα θέματα και άλλες προτεραιότητες στο τέλος θα δείτε ότι τίποτα δεν θα μπορέσει να προχωρήσει. Νομίζω ότι θέσαμε κάποιους κοινού ε, στόχους που είναι να δείξουμε πραγματικά ότι θέλουμε να φτάσουμε σε αποτελέσματα, απτά αποτελέσματα για τους πολίτες που ζουν στην Ευρώπη στα πλαίσια της στρατηγικής για το 2020 και έχω την εντύπωση ότι εδώ η επιλογή είναι απαραίτητη. Μπορεί να είναι δύσκολη, αλλά πρέπει να επιλέξουμε μεταξύ όλων των απαραίτητων θεμάτων κάποιες προτεραιότητες. Δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε όλες τις ανάγκες. Γι' αυτό και θεωρώ ότι θα πρέπει να δούμε βεβαίως τι ενδιαφέρει τους ψηφοφόρους μας, την εκλογική μας περιφέρεια, αλλά θα πρέπει να δούμε και λίγο πιο πέρα από αυτήν την εκλογική περιφέρεια. Τις επόμενες εβδομάδες, τους επόμενους μήνες θα πρέπει πολύ συγκεκριμένα λοιπόν να κοιτάξουμε αυτά τα κεντρικά θέματα, αυτές τις προτεραιότητες. Η άλλη πρόταση την οποία θα ήθελα να θίξω είναι ο προγραμματισμός ο οποίος θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει πολλά διαφορετικά ταμεία τα οποία τα συγκεντρώνουμε σε μία συγκεκριμένη προτεραιότητα. Αυτό καταρχήν ξεκινάει βεβαίως από την ιδέα της απλοποίησης. Καταλαβαίνετε όμως ότι παραμένουν στην Ευρώπη πολλά διαφορετικά ταμεία. Αν αυτά θα πρέπει να συγκεντρωθούν, να προσελκυθούν σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα ή σχέδιο, κινδυνεύουμε να πέσουμε στην παγίδα στα σφάλματα τα οποία κατά κάποιο τρόπο θα είναι πάρα πολύ δύσκολο πρώτον να ελεγχθούν και δυσκολεύουν εξαιρετικά και τη διαχείριση των προγραμμάτων. Θα προσπαθήσω λοιπόν εγώ να αποφύγουμε όσο μπορούμε ε, αυτές τις παγίδες, αυτά τα σφάλματα, βελτιώνοντας βεβαίως τη διαχείριση και θα πρέπει πραγματικά να μην συνεχίσουμε στα ίδια ποσοστά σφαλμάτων, δυσκολιών, όπως και στο παρελθόν. Θα ήθελα λοιπόν εδώ να σας παρακαλέσω πραγματικά να το ξανασκεφτείτε. Εμείς από μέρος της Επιτροπής είμαστε ανοιχτοί στον ε, διάλογο και στη συζήτηση. Θα ήθελα επίσης να σας αναφέρω και ένα άλλο σημείο όσον αφορά την απόφαση σας για τα θέματα που αφορούν την οικονομική διαχείριση και τον έλεγχο. Οι δικές μας προτάσεις για τα θέματα αυτά ουσιαστικά οδήγησαν στην διαδικασία της απαλλαγής. Αυτό είναι μια ενίσχυση του συστήματος ελέγχου, των, της διαδικασίας ελέγχου και βεβαίως η, προχά, η προκάτοχός μου είχε πολύ συγκεκριμένη άποψη για το θέμα αυτό, αλλά πιστεύω ότι έχουν ληφθεί πολύ σημαντικά μέτρα και βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια η ανάλυση των στοιχείων των τελευταίων ετών μας δείχνει ότι πραγματικά έπρεπε να ληφθούν αυτά τα μέτρα και ότι πάνε προς τη σωστή κατεύθυνση. Γι' αυτό και εγώ λοιπόν θα σας ζητούσα εδώ να με υποστηρίξετε, να μας υποστηρίξετε. Τελευταίο σημείο, επίσης πάρα πολύ σημαντικό, που θα ήθελα να συμφωνήσουμε. Πρόκειται για τα δημοσιονομικά εργαλεία. Για τον τομέα αυτό Θα ήθελα να πω ότι υπάρχει μια προσπάθεια επέκτασης από τα προϊόντα στις ποσότητες. Τα εργαλεία αυτά επαναλαμβάνω αυτό γιατί για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, θα πρέπει γρήγορα, με γρήγορες διαδικασίες να φτάνουν στον τελικό δικαιούχο, σε αυτόν που τελικά θα πρέπει να υποφεληθεί. Να μην είναι πάρα πολύ μακριά, αν θέλετε, και στο χρόνο ε, θα πρέπει δηλαδή να θέσουμε κάποιες ε, χρονικές προθεσμίες, όρια, πολύ συγκεκριμένα, έτσι ώστε να μπορεί ο τελικός αποδέκτης να βλέπει το τέλος της διαδικασίας. Το θέμα της καλύτερης ε, και πιο αποτελεσματικής δαπάνης αλλά αυτό με κάποια χρονική, αν θέλετε, ε, ένα χρονικό όριο. Είμαι ανοιχτό και εδώ σε οποιαδήποτε πρόταση, αλλά ξέρετε ότι και εδώ μπορούμε να αλλάξουμε τις προτάσεις μας, είμαι διατεθειμένος να φτάσω μέχρι και στο 1 τρίτο του τελικού ποσού, εάν αυτό δεν έχει ε, δαπανηθεί στο τέλος της προκαθορισμένης περίοδου, να βρεθεί δηλαδή ε, μία λύση. Αλλά πιστεύω ότι εδώ πραγματικά και η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να συμφωνήσουν. Και δεν πρέπει να είμαστε αφελείς από πολιτικής απόψεως όσον αφορά το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Δεν μπορούμε να γνωρίσουμε δηλαδή αυτά που συζητούνται και τη διαπραγμάτευση που λαμβάνει η χώρα εκεί. Η Επιτροπή σας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχει πολύ συγκεκριμένες θέσεις και προτάσεις, αλλά καταλαβαίνετε ότι η Επιτροπή σας δεν μπορεί να αγνοεί την γενικότερη πρόταση που έχει κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο περικοπές υπάρχουν. Απ' την άλλη μεριά θα πρέπει να διασφαλίσουμε την ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και το 2013, όπως ξέρετε, οι μισές χώρες θα χρησιμοποιήσουν 50% τον, ε, θα χρησιμοποιήσουν για τις επενδύσεις τους. Το 50% των ποσών αυτών θα προέρχονται από τα ταμεία και πολλές χώρες πάνω από 60% των επενδύσεων τους θα προέρχεται από τα διαρθρωτικά ταμεία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι οι επιπτώσεις είναι άμεσες και στις διαπραγματεύσεις, στις συζητήσεις που έχουμε, δεν πρέπει να τα ξεχνάμε αυτά. Η Ευρώπη, η στρατηγική για την Ευρώπη του 2020 θέτει συγκεκριμένους στόχους, τα περιφερειακά κονδύλια θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για αυτούς τους συγκεκριμένους στόχους που έχουν τεθεί στη στρατηγική του 2020 και οι 271 περιφέρειες της Ευρώπης θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά αυτά τα περιφερειακά κονδύλια με σκοπό να μειωθούν οι σημαντικές διαφορές που συνεχίζουν να υπάρχουν, λαμβάνοντας υπόψη όμως το γενικό αρχιτεκτόνημα της χρηματοδότησης, την κατανομή που έχει αποφασιστεί, οι περικοπές είναι κάτι που σε πολλές περιπτώσεις είναι αναπόφευκτες Διαβάσατε τις δηλώσεις της Προεδρίας της Κύπρου. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να συνειδητοποιήσουμε ότι οι περικοπές πλήττουν όλες τις πολιτικές και στο εσωτερικό της περιφερειακής πολιτικής αν υπάρξουν συγκεκριμένες περικοπές θα πρέπει να υπάρχει μια ίση αν θέλετε ε, αντιμετώπιση και δεν θα πρέπει κάποιοι να πληρώσουν τα σπασμένα αυτών των περικοπών. Θα ήθελα επίσης ευχαριστήσω για άλλη μια φορά όλους σας για την εργασία σας, τις προσπάθειές σας τους τελευταίους μήνες, τις εκατοντάδες των ε, προτάσεων, συμπληρωματικές τροπολογίες που προετοιμάσατε. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τους εισηγητές για τις προτάσεις τους. Δεν είναι εύκολο. Και θα ήθελα επίσης να σας πω ότι είναι σημαντικό να συνεχιστεί η συζήτηση. Ξεκινάει η τριμερής συζήτηση, διαπραγμάτευση και καταρχήν θα ήθελα να σας πω ότι ως προς την ουσία νομίζω ότι βρισκόμαστε στην σωστή κατεύθυνση και συμβαδίζουμε. Κύριε Επίτροπε, ευχαριστώ πολύ. Να ποιοι θέλουν να πάρουν το λόγο. Κανείς? Α, τότε βλέπω ότι κάποιοι θέλουν. Να ξεκινήσουμε τους συντονιστές και την πρόεδρη. Να κάνουμε κάποιες εξαιρέσεις καμιά φορά, έτσι. Ο Νίκος θέλει πρώτα απ' όλα να πάρει το λόγο. Παρακαλώ, κύριε Χρυσόγελε. Ε, κύριε Επίτροπε, ευχαριστούμε που είσαστε εδώ για να συζητήσουμε. Ήθελα να επισημάνω ε, τέσσερα θέματα. Ε, το ένα που είναι νομίζω πάρα πολύ σημαντικό και ιδιαίτερα αυτή την περίοδο της οικονομικής κρίσης είναι, όπως είπατε και εσείς, να φτάνουν τα χρήματα γρήγορα και να παράγεται αποτέλεσμα ε, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ε, αυτό παρατηρούμε τώρα στην Ελλάδα και επειδή είναι και ένα θέμα με το οποίο νομίζω ασχολείστε, είναι ότι τα χρήματα που είναι διαθέσιμα δεν φτάνουν τελικά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γιατί συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε το θέμα με παλιούς όρους. Δηλαδή, οι τράπεζες όταν αξιολογούν τα προγράμματα μικρομεσαίων επιχειρήσεων, κοιτάνε αν είναι βιώσιμες, βέβαια όλες σήμερα αντιμετωπίζουν προβλήματα, άρα το 80% των αιτήσεων απορρίπτονται. Και όταν υπάρχει, εγκρίνεται το 20%, αυτές οι μικρομεσαίες δεν ξεκινάνε τα προγράμματα, γιατί παίρνουν τα χρήματα μετά από ένα ή δύο χρόνια και πρέπει να έχουν καταβάλει και το ποσό συν το ΦΠΑ που δεν είναι πλέξιμο. Άρα σημαίνει ότι πρέπει σαν Ευρωπαϊκή Ένωση να αλλάξουμε λίγο τη διαδικασία. Αλλιώ δεν έχει νόημα, δεν πρόκειται ποτέ να προωθούν τα χρήματα σε μια περίοδο κρίση. Και είναι πολύ σημαντικό, ακόμα και τώρα οι μικρομεσαίε δεν έχουν δυνατότητα, παράδειγμα, να προμηθευτούν πρώτε ύλε για τι δραστηριότητέ του. Το δεύτερο είναι ένα θέμα που αφορά την περίοδο 14-20 και το έχουμε στήσει πολλέ φορέ και στην Επιτροπή μα τα στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν για να γίνει κατηγοριοποίηση των περιφερειών σε αναπτυγμένες, σε λιγότερο αναπτυγμένες και σε υπομετάβαση. Εάν δεν ληφθούν υπόψη τα πιο πρόσφατα στοιχεία, όσο πιο κοντά στο 2014, υπάρχει ο κίνδυνος η κατάταξη των περιφερειών να γίνει με παλιά στοιχεία, δηλαδή στοιχεία του 9 ή του 10, που είναι είτε πριν της κρίσης, είτε στο ξεκίνημα της κρίσης. Και αυτό θα αλλάξει την ταξινόμηση, το ranking των περιφερειών. Για παράδειγμα, και με βάση μια ε, έκθεση που είχαμε συζητήσει εδώ, όταν εξετάστηκαν στοιχεία, με στοιχεία του 9 η κατάταξη των περιφερειών, ήδη κάποιες περιφέρειες 9 έχουν αλλάξει κατηγορία λόγω ακριβώς των, της κρίσης που επηρεάζει τα, το ΑΕΠ τους. Το τρίτο, το οποίο είναι επίσης νομίζω ιδιαίτερα σημαντικό και επειδή είμαι και εκλεγμένος περιφερειακός σύμβουλος θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι στην επόμενη προγραμματική περίοδο ο ρόλος των περιφερειών είναι αναβαθμισμένος. Όταν μιλάμε για περιφερειακή ανάπτυξη, οι περιφέρειες πρέπει να είναι αυτοί που θα συνυπογράψουν το, το συμβόλαιο εταιρική σχέσης, το contract partnership και να μην είναι απλώς το κράτος μέλος και οι κομισιόν που θα αφασίσουν και για τα περιφερειακά προγράμματα. Δηλαδή, όταν μιλάμε για ένα περιφερειακό πρόγραμμα σε μια περιφέρεια, πρέπει να υπάρχει σύμφωνη γνώμη και του Περιφερειακού Συμβουλίου των Περιφερειακών Αρχών και να έχει γίνει διαβούλευση, ώστε να μην συνεχίζεται αυτό που γίνεται μέχρι τώρα, τα κεντρικά, η κεντρική διοίκηση, ο κράτο αποφασίζει για τι περιφέρειες χωρί τη συμμετοχή των περιφερειών. Δεν υπάρχει περιφερειακή ανάπτυξη αν δεν συμμετέχουν και οι περιφέρειες. Και το τέταρτο που είναι βέβαια ένα γενικότερο θέμα είναι το θέμα των περικοπών. Σε μια εποχή που υπάρχει κρίση πρέπει να αυξηθούν οι χρηματοδοτήσει και το ζητάει το Κοινοβούλιο γιατί δεν μπορεί όλες αυτές οι πολιτικές περιοριστικές να αντιμετωπίσουν τα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα που δημιουργούνται σήμερα. Δηλαδή, στην πραγματικότητα θα έπρεπε να δώσουμε έμφαση στους ιδίους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να βρεθούν δηλαδή περισσότεροι ήδη πόροι, αντί να επικεντρώνουμε στις περικοπές του προϋπολογισμού. Αν δηλαδή το MFF έχουμε λιγότερους πόρους σε μια περίοδο που χρειάζονται περισσότεροι δημόσιοι πόροι και προφανώς και περισσότεροι ιδιωτικοί πόροι, τότε πάμε σε λάθος κατεύθυνση. Και αυτό φαίνεται και στις χώρες κρίση όπως είναι η Ελλάδα, που τα περιοριστικά μέτρα έχουν οδηγήσει και σε διάλυση της οικονομίας και βέβαια και την αποσύνθεση τη κοινωνία. Ευχαριστώ πολύ. Ο κ. Βανίστα ελπίζω Λεμπέρ, να δώσει σας πούμε το παράδειγμα ευσύνων του λόγου. Ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ καλό να αισθάνεσαι πως είναι η ατμόσφαιρα μετά την ψηφοφορία. Να επισημάνω εντάχει τι συνέβη σήμερα το πρωί. Σήμερα εδώ είχαμε μια ψηφοφορία για την πολιτική, κοινή πολιτική αλληλείας. Στα μείζωνα σημεία είχαμε 20 υπέρ 19 κατά ή το αντίστροφο. Πώς είναι τα ψάρια που κολυμπάνε προς κάθε κατεύθυνση. Στην προετοιμασία μας λοιπόν τι κάναμε κι εμείς. Ξεκινήσαμε με βάση μία μακρά συνεργασία με την Κομισιόν και τους ηγητές, τους δονηστές, να επιλέξουμε την κατεύθυνση. Και έτσι μπήκαμε σε μια διαδικασία, εγώ, η Κωνσταντζα και άλλες ηγητές, να επιλέξουμε τα 10 πιο σημαντικά σημεία και εκεί να εστιάσουμε τη συζήτηση για να προχωρήσουμε. Οπότε μπορεί να μην συμφωνούμε 100% στα πάντα, αλλά τουλάχιστον μπορούμε να βρούμε μια κοινή πορεία. Σε σχέση με τα θέματα που εσείς χαρακτηρίσετε ως μίζωνα, να πω και εγώ ότι καταγράφω το εξής. Λοιπόν, να είμαστε σαφείς. Θέλουμε να διαφυλάξουμε την ολοκληρωμένη προσέγγιση. Θέλουμε να έχουμε τις κατάλληλες υποχρεώσεις ώστε να μπορέσει να είναι ομαλή η μετάβαση. Ξέρετε, από την πλευρά όμως υπάρχει και η ευελιξία. Η ευελιξία, όλο και περισσότερη ευελιξία στις περιφέρειες για να κάνουν καλύτερες επιλογές. Είναι και αυτό μια λύση. Δεν φεύγουμε καθόλου, δεν ξεφεύγουμε από τον κανόνα και την κατεύθυνση που είναι ε, οι θεματικές ενότητες. Και να ακούμε, έτσι, να με προσοχή τι λένε τα κράτη-μέλη. Να μην θέσουμε ένα αμφιβόλο την γενική προσέγγιση όπως εσείς την παρουσιάσατε. Ένα δεύτερο σχόλιο για αυτά τα νέα καινοτόμα εργαλεία. Με πολύ χαρά διαπιστώνω ότι στον δημοσιονομικό κανονισμό υπάρχει μια ισχυρή θέση πλέον και από κοινού με την Κομισιόν και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων κινούμεθα στην κατεύθυνση. πρέπει να έχουμε μια σαφή εικόνα τι κονδύλια έχουμε και μπορούν να κατευθυνθούν. Να είναι σαφής, ε, σαφή τα χαρακτηριστικά των δικαιούχων και οι δικαιούχοι να έχουν μια σαφή εικόνα του τι μπορούν να περιμένουν ή όχι. Χρειαζόμαστε λοιπόν αυτά τα νέα εργαλεία. Δεν τι είπε προλαλή Τι βλέπουμε σήμερα. Οι τράπεζε δεν κάνουν τίποτα. Στην Ελλάδα δεν κάνουν τίποτα. Λοιπόν, να είμαστε ειλικρινεί. Τα μόνα χρήματα που εισραίουν στην Ελλάδα είναι πολύ συγκεκριμένα από τα Ταμείο περιφερειακή ανάπτυξη. Και αν μου επιτρέπετε και ένα τελευταίο σχόλιο, τι γίνεται στη, στα κράτη-μέλη μας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη φασαρία για αυτή την εταιρική σχέση, για τον αποκεντρωτικό χαρακτήρα που θα πρέπει να έχουν αυτές οι συμβάσεις εταιρικής σχέσης. Είναι πολύ σημαντικό το επόμενο διάστημα, το επόμενο εξάμεινο αν θέλετε, όλα τα κράτη-μέλη θα κληθούν να παρουσιάσουν τα προγράμματά τους. Για να δούμε λοιπόν πώς μπορούμε να συγκεράσουμε αυτές ε, τις ε, τάσεις και σε επίπεδο προγραμματισμού, σχεδιασμού των προγραμμάτων. Πρέπει λοιπόν να κληθούν τα κράτη-μέλη να ξεκινήσουν ήδη να κάνουν δουλειά. Βλέπω ότι ήδη σε κάποια κράτη-μέλη ήδη γίνεται αυτό. Ώστε να μην είναι η συζήτηση θα υπάρξουν ή δεν θα υπάρξουν και τα χρήματα, μα θα υπάρξουν χρήματα από την πολιτική συνοχή για όλες τις περιφερειές. Εντάξει, μπορούμε να μιλήσουμε για νέε κατηγορίες. Ναι, αλλά θα υπάρξουν διαθέσιμα κονδύλια. Οπότε, α καθίσουμε με τους πολίτες, με τους εκπροσώπους των πολιτών, σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Να συζητήσουμε πώς ακριβώς θα λειτουργήσει αυτή η πλέον σημαντική πολιτική επενδύσεων για να μπορέσουμε να έχουμε πραγματική ανάπτυξη και θέσει εργασία. Χαίρομαι ιδιαίτερα με αυτό που λέει η Κομισιόν. Διαπραγμάτευση. Πού είναι το κακό στη διαπραγμάτευση. Ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντζα. Ε, ε, Ευχαριστώ, Ντανούτα. Ευχαριστώ τον Επίτροπο. Και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί Είπατε ότι σε πολλά σημεία βρισκόμαστε πολύ κοντά και έχω την εντύπωση ότι αυτά τα οποία αναφέρετε ως σημεία που συνεχίζουν να δημιουργούν προβλήματα, δυσκολίες, ε, μπορούν να εξελιχθούν από τη στιγμή που οι στόχοι μας είναι κοινοί και από τη στιγμή που οι θέσεις μας μπορούμε να συνεργαστούμε, να συζητήσουμε και να βρεθούμε κοντά. Για μένα ο δύσκολος εταίρος είναι το Συμβούλιο. Εκεί μπορεί να υπάρξουν δυσκολίες και μπορεί τελικά να μην βρεθεί κοινή προσέγγιση. Θα ήθελα να σας αφέρω δύο σημεία. Μιλήσατε για την διευκόλυνση Connecting Europe και συνδέοντας την Ευρώπη. Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί τον Ιούλιο η ψηφοφορία έδειξε με σαφήνεια ότι θέλουμε να φτάσουμε σε έναν συμβιβασμό. Το θέμα βέβαια είναι τώρα αυτά τα 10 δις, ο γενικός κανονισμός, θα δώσει τις πιο συγκεκριμένες κατευθύνσεις και νομίζω ότι εδώ θα πρέπει εσείς με τον κύριο Λάμπερτ, με μένα, να προσπαθήσουμε να βρούμε έναν τρόπο γιατί αυτό που επιθυμεί εδώ το Συμβούλιο είναι να μην τα βρούμε, να υπάρξει μεγάλη αντιπαράθεση και τελικά να μην προχωρήσει αυτή η διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη. Γι' αυτό και θεωρώ ότι θα πρέπει να καταλάβετε ότι και εμείς είμαστε ανοιχτοί σε κάποιες συμβιβαστικέ λύσεις και έχουμε ένα περιθώριο ελιγμού το οποίο θέλουμε να το χρησιμοποιήσουμε. Υπάρχει λοιπόν η ψηφοφορία τον Οκτώβριο, αλλά επειδή όλα δεν συμπεριλαμβάνονται στο γενικό κανονισμό, υπάρχει, επαναλαμβάνω, δυνατότητα περαιτέρω συζήτησης. Δεν νομίζω ότι από τη δική μας πλευρά υπάρχουν σοβαρές ε, δυσκολίες. Η χρησιμοποίηση των νέων ε, δημοσιονομικών εργαλείων είναι πάρα πάρα πολύ ε, σημαντικές και δεν νομίζω ότι εδώ πρέπει να δημιουργήσουμε δύο ομάδες, αυτοί που είναι υπέρ της πολιτικής συνοχής και αυτοί που είναι υπέρ των περικοπών. Υπάρχει ε, δυνατότητα κοινή κατεύθυνσης και συνεργασίας. Κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να μου πείτε και κάτι άλλο η διαπραγμάτευση η δημοσιονομική για το 2012 δημιούργησε δυσκολίες στο θέμα της πολιτικής συνοχής και σαφώς το Συμβούλιο δεν είχε, από ό,τι φαίνεται, τις απαραίτητες προβλέψεις για τις πληρωμές. Θα ήθελα να μου πείτε πώς βλέπετε τα πράγματα για το 2013 υπάρχει περίπτωση να εμποδιστεί η διεξαγωγή προγραμμάτων ακριβώς επειδή θα βρεθούμε αντιμέτωποι με το ίδιο πρόβλημα. Όσον αφορά τις πληρωμές, γιατί άλλο είναι να μην εγκριθεί ένα πρόγραμμα, άλλο είναι μία περιφέρεια να μην μπορεί, να μην είναι σε θέση να υλοποιήσει ένα πρόγραμμα και άλλο είναι να μην φτάνουν οι πληρωμές και αυτό να οφείλεται καθαρά στο Συμβούλιο. Ευχαριστώ, Ραμόνα Μανέσκο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να συγχαρώ τον Επίτροπο για την παρουσίασή του και δεν θέλω να επαναλάβω τα όσα έχουν ήδη αναφερθεί. να ε, βασιστώ μόνο σε αυτό που είπε η συνάδελφος προηγουμένως για τις περιφέρειες και για τα προγράμματα και έργα που έχουν εγκριθεί και δεν έχουν υλοποιηθεί. Μπορώ να σας αναφέρω συγκεκριμένα το Εράσμους για τους ε, τοπικούς εκπροσώπους. Είναι κρίμα που ακόμα Μιλάμε για στήριξη του τοπικού και περιφερειακού επίπεδου, αλλά στην πράξη δεν καταφέρνουμε να υλοποιήσουμε ε, τα όσα αποφασίζουμε και είναι κρίμα που δεν έχουμε καταφέρει να το υλοποιήσουμε αυτό το πρόγραμμα ε, όπως πρέπει, παρόλο που οι περιφέρειες έχουν υποβάλει προτάσεις και έχουν ε, αναπτύξει προγράμματα. Μπορείτε να μας εξηγήσετε κύριε Επίτροπε πότε θα ολοκληρωθεί και θα υλοποιηθεί αυτό το project που είναι πολύ χρήσιμο για τις κοινωνίες. Ευχαριστώ. Αλφονσί. Θα απαντήσει ο Επίτροπος βεβαίως ε, σε όλα τα ερωτήματα, ιδίως για το ε, δημοσιονομικό πλαίσιο, γιατί βεβαίως είναι ε, σημαντικό το θέμα, μεγάλη πρόκληση. Θα μπορούσε ακόμα να οδηγήσει και σε ακύρωση του διακτημένου της πολιτικής συνέχεια της Ευρώπης παρόλο που υπάρχει αλληλεγγύη βεβαίω μεταξύ Επιτροπή και Κοινοβουλίου, πρέπει κάποια στιγμή να καθορίσουμε ένα κατόφλι κάτω από το οποίο τα πάντα αμφισβητούνται και θέτονται αναφιβόλω. Θα πρέπει λοιπόν να αναλάβουμε όλε τι ευθύνε μα. Ευχαριστώ, Ολτζι Βλάσακ. Ευχαριστώ. Χαίρομαι ιδιαίτερω που είμαστε σε θέση να συζητήσουμε μαζί σας ε, την πολιτική συνοχή. Θα ήθελα να επαναλάβω αυτά που είπε η κυρία Κράμολ στις παρατηρήσεις σας, γιατί υπάρχει ένας μεγάλος κίνδυνος εδώ. Ε, και σας παραπέμπω στην συζήτηση εδώ χθε με τον Επίτροπο Κάλλας, όπου δυστυχώς δεν ήταν ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη η στάση του σε ό,τι αφορά τι δικέ μα απόψει και ανάγκε. Γι' αυτό θα ήθελα να πιστήσω την προσοχή σα ε, στι προτεραιότητέ μα, δηλαδή στην ενίσχυση του ρόλου των τοπικών και περιφερειακών αρχών και των ε, φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης στη διαδικασία βελτίωσης ε, αυτού, αυτής της σύμβασης Θεωρώ ότι οι κυβερνήσεις θα πρέπει να προετοιμάσουν καλά αυτή την, ε, την σύμβαση τρικής σχέσης. Τώρα, σε ό,τι αφορά την εδαφική διάσταση και το ε, μέσο ITI, παρόλο που βεβαίως ε, ανοίγουμε πλώρη σε, σε νέα νερά, ε, η εδαφική διάσταση, ωστόσο, εκεί δεν έχει λάβει την επαρκή στήριξη. Γι' αυτό ε, θα βασιστούμε σε μεγάλο βαθμό στι αποφάσει που θα ληφθούν τα κράτη-μέλη. Θεωρείτε ότι θα ήταν καλό να ε, εκδοθούν συστάσεις προς τα κράτη-μέλη από την Επιτροπή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριο Μαζί. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, δεν θέλω να ε, είμαστε αποσιόδοξοι, αλλά πρέπει να ανησυχούμε και για την περιφερειακή πολιτική. Έχουμε την αίσθηση ότι το, τα ταμεία συνεχής, τα διαφορετικά ταμεία ε, έχουν χάσει τον αρχικό τους ρόλο, ουσιαστικά είναι ένας μεγάλος κουμπαράς ε, όπου πηγαίνει ο καθένας για να χρηματοδοτήσει άλλες, ε, άλλα προγράμματα με άλλους στόχους. Ε, υπάρχουν παραδείγματα που συζητήσαμε και χθε, όπω ε, τα 10 δι ε, για τον μηχανισμό διασύνδεση. Είναι βασικό, είναι σημαντικό αυτές ε, οι αρχές να διατηρηθούν ακόμα και κατά την εφαρμογή αυτών και την αξιοποίηση αυτών των 10 δι. Άλλο ερώτημα αφορά την αξιοποίηση των ελευθερωτικών ταμείων για την χρηματοδότηση της ε, πολιτικής ανάπτυξης. Δεν είναι κάτι καινούριο. Ε, συμβαίνει συχνά ε, να μην υπάρξει σωστή κατανομή αυτών των κονδυλίων και γι' αυτό είναι σημαντικό να υπάρχουν εχέγγυα ε, για την ε, σωστή αξιοποίηση αυτών των κονδυλίων, ότι οι στόχοι της περιφερειακής πολιτικής θα γίνουν σεβαστοί. Ε, για να επιτύχουμε τα όσα έχουμε θέσει ως στόχους. Ε, τρίτον, δεν ξέρω αν κάνω λάθος, έχω την αίσθηση ότι η κοινή γεωργική πολιτική λαμβάνει κεντρικό ρόλο. Δεν ξέρω βέβαια αν θα υπάρξει σημαντική μείωση των ε, κονδυλίων σε ό,τι αφορά την κοινή γεωργική πολιτική αλλά ε, από ό,τι κατάλαβα περνάμε ε, σε σημαντικές ε, περικοπές στον προπολογισμό σε ό,τι αφορά την περιφερειακή πολιτική. Και εδώ θεωρώ ότι υπάρχει πολιτική επιλογή. Δεν την αποδέχομαι εγώ ως μέλος αυτής της Επιτροπής. Ευχαριστώ. Κύριε Πετρούμα, θέλετε να απαντήσετε. Μάλιστα. Αν δεν απαντήσω σε κάποια από τα ερωτήματα, δεν σημαίνει ότι αναγκαστικά διαφωνώ. Να δούμε τη σειρά τα ερωτήματα για την ε, οικονομική μηχανική, ναι, κατανοώ ακριβώς τη στάση που έχετε ακολουθήσει το τελευταίο διάστημα και, και αυτά που έχετε εγκρίνει και στο οποίο έχετε συμφωνήσει και γι' αυτό, για παράδειγμα, τα κεφαλαία κινδύνου πλέον χρησιμοποιούνται και άρα το, το δεν είναι μόνο να συμφωνούμε στη θεωρία για τα ταμεία, αλλά τα κονδύλια να φτάνουν στον τελικό δικαιούχο. Κάναμε ήδη προτάσεις ε, για την ε, α, κείμενη δημοσιονομική περίοδο. Ξέρω ότι κάποιες φορές υπάρχουν καθυστερήσεις. Ε, κάποιες φορές είναι πολύ αργά ήδη να διαπραγματευτούμε τα σκαντάδες συμβάσεις που ήδη έχουν υπογραφεί, αλλά για την επόμενη περίοδο θα πρέπει να εγγυηθούμε α, ότι δεν θα λειτουργήσει το το σύστημα τον ίδιο τρόπο, ώστε να μην μπορεί να μην έχει πρόσβαση ο δικαιούχος ε, στα ποσά. Αριθμητικά ποσά. Πάντοτε μιλάμε για ε, τελευταία διαθέσιμα στοιχεία που συνήθως η, τα δημοσιεύει γύρω στο Φλεβάρι-Μάρτι. Αν μιλάμε για περιφερειακό επίπεδο πάμε ε, σε ορίζοντα δύο ετών πίσω. Και αν μιλάμε για εθνικά στοιχεία, παίρνουμε ως περίοδο αναφορά στο προηγούμενο έτος. Και τα διεθνωτικά ταμεία παίρνουμε τον μέσο όρο των τελευταίων τριών διαθέσιμων ετών. Αυτή είναι η διαδικασία που ακολουθούμε. σε ό,τι αφορά δηλαδή τη χρήση αριθμητικών στοιχείων και τι σημαίνουν αυτά. Ε, αν εφαρμόσουμε τα στοιχεία μόνο για την επόμενη χρονιά, αυτό θα έχει πολύ μικρό αντίκτυπο. Ε, Ούτω ή δεν περιμένουμε σημαντικέ αλλαγέ από τώρα έω την επόμενη χρονιά στην Ελλάδα. Αν δηλαδή συγκρίνουμε το 2012 με το 2013 μιλάμε για τη σχέση περιφερειών. Συνολικά, ναι, μπορεί το ΑΕΠ να δείξει χαμηλότερα επίπεδα. Διακυβέρνηση σε πολλαπλά επίπεδα και συμμετοχή των περιφερειών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει πρώτα απ' όλα να σέβεται ε, τους συνταγματικούς περιορισμούς των κρατών μελών. Δεν μπορούμε δηλαδή να παρεμβαίνουμε σε τέτοια ζητήματα. Ήδη όμως υπάρχει ένα άρθρο για την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. Θέλω και πάλι όμως να σας καθησυχάσω ότι εμείς παρακολουθούμε πώς τηρείται αυτό το άρθρο και πώς το τα κράτη-μέλη το σέβονται στην πράξη. Θα δούμε λοιπόν με ποιο τρόπο οι περιφέρειες, αλλά και σε τοπικό επίπεδο και αν κρίνεται αναγκαίο, οι μη κυβερνήσεις οργανώσεις συμμετέχουν στην υλοποίηση των επικρισιακών προγραμμάτων και των ε, συμβάσεων ε, εταιρικής σχέσης. Για τα υπόλοιπα που είπατε, εγώ συμφωνώ απόλυτα και συμμερίζομαι τις θέσεις σας. Σε ό,τι αφορά αυτά λεγόμενα του Λάμπερτ. η θεματική συγκέντρωση και η ολοκληρωμένη προσέγγιση δεν είναι οξύμορο σχήμα. Αυτό που προτείνουμε εμείς, αν θέλετε, είναι ένα μενού. Μενού τριών πιάτων. Γιατί θεωρούμε ότι αυτό είναι πιο γήινο από ότι ένα μενού έξι πιάτων. και υπάρχει επαρκή ευελιξία και ελευθερία στις περιφέρειες να επιλέξουν. Μπορεί να είναι πρόκληση η δυνατότητα επιλογή, αλλά πάντοτε πρέπει στην πολιτική ζωή, στον πολιτικό βίο, να υπάρχει η πρόκληση των επιλογών. Οπότε, από το να έχεις έξι διαφορετικούς στόχους που να καλύπτουν όλα τα συμφέροντα σε μια περιφέρεια, μπορεί να σας φαίνεται καλύτερο. Αλλά τελικά, με αυτόν τον τρόπο, αποδυναμώνεται αν θέλετε, η όλη ιδέα που κρύβεται πίσω από την ε, θεματική συγκέντρωση. Φυσικά θα πρέπει να υπάρχουν θεματικοί στόχοι και θα πρέπει να ευθύνη των περιφερειών και των κρατών μελών να επιλέξουν. Είναι αναπόφευκτο κατά τη γνώμη μας αυτό. Σε ό,τι αφορά τη διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη, τα έχουμε πει νομίζω ήδη όλα. Εγώ, ως Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής, μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχω προσωπικό ενδιαφέρον να βρεθεί κατάλληλη λύση. Διότι όλη η ιδέα αυτής της διευκόλυνσης είναι κάτι που συμμερίζεται η μεγάλη πλειοψηφία και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο και εκτός θεσμικών οργάνων, άρα πρέπει να βρούμε μια λύση για να διασκεδάσουμε τις κάποιες ανησυχίες. Όμως αυτό είναι εφικτό θεωρώ. Σε ό,τι αφορά τις πληρωμές, πράγματι, έχουμε μεταφέρει πολύ σημαντικά ποσά σε επίπεδο, επίπεδο δις. Έχει γίνει μεταφορά σημαντικών ποσών από πέρυσι στη φετινή χρονιά. Οι πληρωμές ε, του 2012 ξεκίνησαν μόλις τον Απρίλιο. Το πρώτο τρίμηνο ουσιαστικά αφορά πληρωμές του προηγούμενου έτους. Σύμφωνα με τον προπολογισμό που έχουμε στη διάθεσή μας, είναι τεράστια η πιθανότητα να αυξηθεί αυτός ο όγκος ε, χρημάτων που θα πρέπει να μεταφέρεται και αν δεν υπάρξει πρόσθετος προπολογισμό για φέτος, ίσως τελικά να πρέπει να μεταφέρουμε πάλι, ποσά να κάνουμε carry over ε, κάποιων μικρών διψήφιων ποσών σε δισεκατομμύρια, λέει ο μιλητής, για την επόμενη χρονιά. Μπορεί λοιπόν κάποια project τελικά να κινδυνεύσουν. Αυτό είναι αλήθεια διότι προχρηματοδοτείται τρόπον την προπολογισμό. Οπότε όσο αργεί η επιστροφή των χρημάτων, το, για μεγαλύτερο διάστημα θα πρέπει να εξυπηρετείς το δάνειο που έχεις πάρει. Άρα υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Οπότε αυτό θα αναγκάσει τα κρατημέλη να ε, εμείνουν στη συμφωνία που είχαμε τις προηγούμενες χρονιές. Και το άλλους είναι ειδικά τους τα κορνδύλια. Τώρα το Erasmus για, σε τοπικό επίπεδο, Erasmus for Locals. Ε, είναι μια καλή πρωτοβουλία. Έχουμε αντιμετωπίσει δυσκολίες, αλλά συμφωνήσαμε με την Επιτροπή των Περιφερειών επίσης να έχουμε μια βαθμιαία προσέγγιση. Και την επόμενη χρονιά ελπίζω να ξεκινήσουν οι πρώτες δραστηριότητες που θα εμπλέκουν ε, τους ε, ε, εκπροσώπους ε, σε τοπικό επίπεδο, τους δημοσίους υπαλλήλους ε, σε τοπικό επίπεδο να έχουν ανταλλαγές απόψεων για αυτά τα ζητήματα. Σε ό,τι αφορά τις συμβάσεις εταιρικών σχέσεων, νομίζω τα είπαμε, η εδαφική διάσταση, τα ITI, δεν υπάρχουν συγκεκριμένες διατάξεις ε, πρόνοιες για τα κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη και οι αστικές δομές που έχουν θα αποφασίσουν πώς θα χρησιμοποιήσουν τα χρήματα όσο γίνεται πιο ολοκληρωμένα. Ευχαριστώ. Thank you. Colleagues, I would Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Θέλω να κλείσω τον κατάλογο των ε, αγορητών. Οχτώ αγορητές ακόμη στον κατάλογο. Παρακαλώ να κλείσουμε το κατάλογο και να περιοριστείτε στα τρία λεπτά έκαστος για να έχει άλλα 15 λεπτά ο Επίτροπος. Ο κύριος Σέιρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, στην πρόταση κανονισμού για την εδαφική συνεργασία, η Επιτροπή δεν περίλαβε καμία μνήμα σε ό,τι αφορά τις παραμεθόριες περιφέρειες να είναι επιλέξιμες σε αυτά τα προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας. Αντίθετα, και σε σχέση με ό,τι μας είχατε πει σε μια άλλη συνάντηση που είχαμε στο Στρασβούργο, μαζί με τους ευρωβουλευτές από τις παραμεθόριες περιφέρειες. Γιατί λοιπόν γίνεται αυτή η εξαίρεση για αυτές τις παραμεθόριες ε, περιφέρειες. Γιατί έχουμε το κριτήριο των 150 χιλιόμετρων. Ξέρετε, οι πορτογαλικές περιφέρειες και οι Αζόρες συγκεκριμένε, γνωρίζετε κύριε Επίτροπε, ότι αυτόματα αποκλείονται οι πορτογαλικές περιφέρειες για την επόμενη δημοσιονομική περίοδο. Και άρα η πολύ σημαντική διάσταση δευτερική συνεργασίας που είναι αυτή ακριβώς, γιατί είναι πολύ σημαντικό κομμάτι ε, της χρηματοδότησης που λαμβάνουν. Και τι συμβαίνει λοιπόν με την πρότασή σας ακολούθησα η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μελλοντική στρατηγική για τις παραμεθόριες ε, περιφέρειες, όπου αναφέρεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ανοιχτή για να διευκολύνει την ε, διασυνοριακή συνεργασία των παραμεθόρων περιφερειών, αρκεί ε, η, η απόστασή τους από τις ακτές να είναι 150 χιλιόμετρα. Άρα, σε αντίθεση λοιπόν με αυτό που προβλέπει η ανακοίνωσή σας, που δηλαδή θέλετε να διευκολύνετε αυτή τη συνεργασία, δεν βλέπουμε όμως τίποτα πρακτικά στην πρόταση. Θα θέλαμε κάποια διευκρίνηση, κύριε Επίτροπε, επ' αυτού. Γιατί εδώ βλέπω πραγματικά μια ανακολουθία ανάμεσα στα δύο έγγραφα. Στις 14 Αυγούστου μάλιστα λάβουμε μια απάντησή σα που λέει το εξή. Θα τη διαβάσω. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ανοιχτή να διευκολύνει τη διασυνοριακή συνεργασία των παραμεθόρων περιοχών ε, σε ό,τι αφορά τα θαλάσσια σύνορα όταν ξεπέρνουν τα 150 χιλιόμετρα από την ακτή αλλά δεν κρίνει αναγκαία οποιαδήποτε πρόταση τροποποίησης της αρχικής της πρότασης. Άρα, ρωτώ, πώς είναι δυνατόν από τη μία σε ένα μεταγενέστερο έγγραφο από την ομοθετική σας πρόταση, δηλαδή να φέρουμε στην ανακοίνωση, να λέτε ότι είσαστε ανοιχτοί να αναξαναδείτε, να αναθεωρήσετε αυτό το ζήτημα, ώστε να υπάρχει μια καλύτερη διεθνική συνεργασία για τι παραπεθόρε και νησιωτικέ περιοχέ. Και τώρα, μετά στη γραπτή σα απάντηση, τι μου λέτε. Ναι, ναι, ναι, διευκολύνουμε, αλλά δεν υπάρχει κανένα λόγο να τροποποιήσουμε ε, την νομοθετική πρόταση. Κοιτάξτε. Ε, το πορτογαλικό δίκαιο υπάρχει μία έννοια που είναι η της διανοητικής επιφύλαξης. Δηλαδή δεν μπορούμε άλλα να λέμε και άλλα να κάνουμε να σας το πω έτσι πολύ συνοπτικά. Εδώ βλέπω μια πρακτική ανακολουθία. Άλλα λέτε, άλλα κάνετε. Ε, δεν είναι δυνατόν μία στιγμή να λέτε όχι, όχι, δεν πρόκειται να διευκολύνουμε αυτή την εργασία και το βλέπουμε στην πράξη και από την άλλη στην ανακοίνωσή σας για το μέλλον των παραθύρων περιφερειών και λέτε είμαστε ανοιχτοί να το ξαναδούμε. Και μετά στην γραπτή απάντηση που μου δίνετε πάλι μου λέτε όχι, δεν βλέπουμε ότι είναι αναγκαίο να γίνει κάτι τέτοιο. Ε, συνεχώς βλέπω να αλλάζετε θέση. Δεν κατανοώ αυτή τη στάση και θα ήθελα κύριε Επίτροπε να μου εξηγήσετε ε, και να μου σχολιάσετε αυτό το γεγονός. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Όλπριχτ. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονό ότι η Επιτροπή μόλι τώρα έχει ξεκινήσει τι διαπραγματεύσει με τον τριμερή διάλογο, γιατί Όταν μας παρουσιάσατε τις απόψεις σας για το συμβιβασμό του Κοινοβουλίου, μας ενημερώσετε για το ποια θα είναι η θέση της Επιτροπής της Διαπραγματεύσης. Αυτό θα μας είναι πολύ χρήσιμο στο μέλλον. Γιατί έχουμε ένα περιθώριο λιγμών ε, και από τις δύο πλευρές. Ας περάσω τώρα στα πιο συγκεκριμένα. Βεβαίως, ε, σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Ε, είμαστε σίγουροι και θεωρούμε δεδομένο ότι θα κάνετε ό,τι είναι δυνατόν. Το θέμα είναι βέβαια τι είναι δυνατόν να γίνει. Σε ό,τι αφορά τις προτεραιότητες, τα διασυνοριακά έργα, όλα εντάξει. Το μόνο στοιχείο για μας είναι η μέθοδος. Και είμαστε τεθειμένοι να καταλήξουμε σε συμβιβασμό, ε, αρκεί να λαμβάνονται υπόψη και τα και τα εθνικά κονδύλια. Και αυτό είναι τμήμα της ε, πολιτική συνοχής. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα λοιπόν με τους στόχους, αλλά σε ό,τι αφορά τη μέθοδο δεν είναι δυνατόν να τα αφαιρέσουμε από τα εθνικά κονδύλια, τουλάχιστον όχι στην αρχή, ίσως στη συνέχεια. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να καταλήξουμε σε συμβιβασμό. Σας μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι δεν περιμένουμε περιμένουμε και τι θα γίνει και από την πλευρά της Επιτροπής. Δεύτερο στοιχείο. για τις βαριές υποδομές, για τις πιο ανεπτυγμένες περιφέρειες ε, από το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Θα ήθελα ο Επίτροπος να μας ε, δώσει κάποια στοιχεία για το τι απαιτείται για την επίλυση των προβλημάτων. Η Επιτροπή εξ αρχή λέει ότι οι υποδομές για τις βασικές υπηρεσίες ό,τι αφορά ε, τις μεταφορές, το περιβάλλον και το ICT. Πάντα ήταν δύσκολο να, να καταλήξουμε σε ορισμό των βασικών υπηρεσιών. Τι ακριβώς εννοούμε με αυτό τον όρο. γιατί ήδη και έχουμε πρόβλημα και με τις πιο ανεπτυγμένες ε, περιφέρειες. Γιατί το Κοινοβούλιο βεβαίως εκφράζει ε, τις απόψεις ε, των Ευρωπαίων πολιτών. Σε ό,τι αφορά τη θεματική συγκέντρωση, όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να υπάρχει πραγματικά ισχυρή συγκέντρωση, αναμφιβόλως. Τώρα για το κατά πόσο πρέπει να είναι τρει ή έξι, καλύτερα πράγματι να έχουμε τρει. Ακόμα καλύτερα θα ήταν να είχαμε δύο. Αλλά ιδίω εν μέσω κρίση ε, η ευελιξία είναι το παν. Η ευελιξία εντό τη συγκέντρωση. Προσπαθούμε λοιπόν οι τελικοί δικαιούχοι να έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τις προτεραιότητες τους, ε, να εξηγήσουν σαφέστατα γιατί, αλλά με απόλυτη συγκέντρωση, ναι. Το θέμα είναι βεβαίως ποιο είναι το πεδίο αυτού του, αυτής της θεματικής συγκέντρωσης και εκεί είναι και το περιθώριο ελεγμών μας. Αυτή η θεματική συγκέντρωση πρέπει να, να είναι πάνω κάτω ίδια ή παρόμοια στους διαφόρους κανονισμούς. Γιατί έχουμε άλλα στοιχεία στο Ταμείο συνοχή, άλλα στον, ε, στο κανονισμό για την περιφερειακή συνεργασία και το καθεξής. Ίσως ε, μέσα στις διαπραγματεύσεις να βρούμε τρόπο να είναι τουλάχιστον παρόμοιες οι διατάξεις. Τώρα για την σύμβαση εταιρική σχέσης, επειδή το συζητήσαμε και στο Στρασβούργο, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον το γεγονός ότι η σύμβαση εταιρικής σχέσης ε, ε, στο πλαίσιο, βασίζεται σε ε, κονδύλια του Ταμείου Συνοχής. Έχουμε πέντε, αυτό είναι κάτι καινούργιο, γιατί έχουμε πέντε ταμεία. Και προτείνεται να στείλετε ε, τις συμβάσεις συνεργασίας μαζί με τις συμβάσεις σχέσεις ταυτόχρονα. Αυτό σημαίνει και τα προγράμματα γεωργικής συνεργασίας. Γιατί οι συμβάσει σχέσεις είναι πέντε. Έτσι απαιτείται συνεργασία μεταξύ όλων των φορέων. Γιατί τα, οι συμβάσει σχέσεις σχέσει δεν αφορούν μόνο ε, τα, τα, το Ταμείο Συνοχή. Είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή και τελευταίο και πιο δύσκολο ερώτημα, όχι για να επιτεθώ στον Επίτροπο, αλλά για να μας εξηγήσετε. Και αν δεν έχουμε αυτή την ε, συμφωνία και αν δεν έχουμε νομική βάση μετά το 2013, τι θα γίνει με την ε, πολιτική συνοχή. Δεν θέλω να προκαλέσω πολιτικό διάλογο, αλλά ε, πρέπει να φανταστείτε και αυτό το ενδεχόμενο, ιδίω όσοι ασχολούνται με τον προπολογισμό. Τι θα γίνει με την πολιτική συνοχή αν δεν υπάρξει συμφωνία, δεν υπάρξει δημοσιονομικό πλαίσιο. Και τι θα συμβεί τότε λοιπόν. Και η Επιτροπή μας θέλει να το μάθει αυτό. Να έχει και αυτό το αρνητικό ενδεχόμενο κατά νου. Γιατί είναι αρνητικό βεβαίω το να μην υπάρχει η νομική βάση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. ευχαριστώ. Θα αναφερθώ στο θέμα του πολίτου, δημοσιονομικού πλαισίου και αφήστε με να θέσω το θέμα αλλιώς. Θέλετε να παραμείνουμε σαν σκυλάκια υπομονετικά στην ουρά για να δούμε τι θα μας δώσουν, τι θα θελήσουν να μας δώσουν. Μιλάμε από τη μία για την ανάπτυξη, την ανάγκη να καλύψουμε τις ανάγκες ε, των συγκεκριμένων χωρών και από την άλλη ακούμε για περικοπές. Η ερώτησή μου λοιπόν κύριε Επίτροπε είναι πολύ συγκεκριμένη και μία. Τι άλλες δικαιολογίες θα βρείτε να μας δώσετε. Ξέρουμε τις παλιές δικαιολογίες όσον αφορά τις περικοπές. Εγώ ακούω όλους τους επικεφαλείς κρατών και κυβερνήσεων να λένε χρειαζόμαστε χρήματα, χρειαζόμαστε ένα σχέδιο Marshall για την Ευρώπη, χρειαζόμαστε ανάκαμψη και ανάπτυξη και από την άλλη περικοπές. Πού υπάρχει λογική. Πώς μπορούμε λοιπόν να βγούμε από, αυτό το, από αυτήν την κατάσταση. Όπως είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητές. Μιλάμε για κάτι το πάρα πολύ συγκεκριμένο και ρεαλιστικό. Εγώ θέλω να δω πώς θα κινηθεί το Συμβούλιο. Ίσως εσείς ξέρετε εξάλλου, γι' αυτό και σας θέτω αυτή την ερώτηση. Και κάτι άλλο ακόμα. Μακροοικονομικές προϋποθέσεις. Ξέρουμε πολύ καλά αυτά που συζητούμε εδώ μεταξύ Επιτροπής και Κοινοβουλίου. Από την άλλη όμως υπάρχει το Συμβούλιο. Τα πράγματα ποτέ δεν συμβαίνουν όπως θα έπρεπε στο Συμβούλιο. Και όσον αφορά την διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη, δύο πράγματα είναι πολύ σημαντικά. Πρώτον, πώς θα υπάρξει ροή των κονδυλίων πραγματική ροή και δεύτερον να μην βρεθούν οι μικρές χώρες πάλι στην ουρά και να μην υποστούν ένα νέο πλήγμα. Θα σε ευχαριστώ. Ο κύριος Άλβες. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να χαιρετήσω τον Επίτροπο που το προηγούμενο Σαββατοκύριακο ήρθε στην περιφέρειά μου, ε, διέτρεξε διάφορες νήσους και νομίζω ήρθε προετοιμασμένος αυτή τη συνάντηση. Να πω το εξή. Το Συμβούλιο, σε ανακοίνωση του Ιουνίου, επιβεβαίωσε ότι η βασική προτεραιότητα παραμένει ισχυρή, α, βιώσιμη, α, ανάπτυξη για όλους. Όμως μετά ήρθαν οι άλλες ειδήσει ότι το ανώτερο επίπεδο των συνολικών δαπανών για την επόμενη περίοδο θα πρέπει να μειωθεί, ότι θα πρέπει ε, να υπάρξει μια τάση και προσπάθεια περικοπής όλων των κονδυλίων σε όλους τους τομείς και Αναρωτιέμαι, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ε, οι Κομισιόν μπορούν να θέσουν να αμφιβάλλω ε, τα κονδύλια που προορίζονται για τη συνοχή. Μπορείτε να μου σχολιάσετε αυτό, γιατί θυμάμαι πολύ καλά τη στρατηγική της Λισαβόνας. Μια στρατηγική που όριζε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση το 2010 ήδη θα πρέπει να είναι η πιο ανταγωνιστική οικονομία στον κόσμο. Θυμάμαι ότι λόγω ελλείψεων και προβλημάτων. Ήδη το 2010 ζούσαμε ε, τη δινή κρίση που δεν έχουμε ξεπεράσει ακόμη. Ζούμε στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση, αντιμετωπίζουμε τεράστια οικονομικά προβλήματα και οι μακροοικονομικές ισορροπίες που θα θέλαμε να έχουν πετύχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τις έχουμε επιτύχει έχουμε ελλείμματα, δημοσιονομικά ελλείμματα, τα οποία τρέχουμε να, θέλετε να σώσουμε και να διορθώσουμε α, ε, συνεχώς. Η πολιτική συνοχή όμως δεν είναι ακρογωνίως λήθος για την ε, οικοδόμηση της νέας Ευρώπης. Είναι κάτι που μπορεί να τεθεί ένα αμφιβόλο, αναρωτιέμαι. Και σύμφωνα με όσα μας είπατε εσείς, ε, και συμφωνώ και επαυξάνω, είναι ότι οι περιφέρειες είναι πάρα πολύ σημαντικές ε, για το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Όμως ε, ταυτόχρονα ε, ισχύει και κάτι άλλο. Ότι οτιδήποτε είναι καλό για τις περιφέρειες είναι καλό για την Ευρώπη εν γέννη. Θα ήθελα λοιπόν να αναφερθώ στον μηχανισμό διασύνδεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα έχει ως σκοπό να φέρει πιο κοντά τις πλέον απομακρυσμένες περιφέρειες. Όμως τελικά φαίνονται αυτές να αποκλείονται. Τι μπορεί να γίνει πρακτικά γι' αυτό. Μία Ματσόνη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για την παρουσία σας στη Επιτροπή μας σήμερα. Σε ό,τι αφορά τη μέθοδο εργασίας για το μέλλον, αναρωτιέμαι Μήπως είναι σκόπιμο να συμφωνήσουμε με βάση το πρόγραμμα του περασμένου Ιουλίου να προχωρήσουμε με θεματικές ενότητες, ώστε στις συναντήσεις μας να συμμετέχουν όλοι οι σχετικοί εισηγητές ανακανονισμό και να μην κατακαιρματίζουμε τελικά, αν κατάλαβα καλά τελικά, αυτή είναι, αυτός είναι ο προσανατολισμός τώρα, να κατακαιρματίζουμε τη συζήτηση ανακανονισμό διότι ο γενικός κανονισμός είναι αυτός που βεβαίως εμπνέει και το περιεχόμενο των τομιακών κανονισμών. Και όπως έγινε και με τις τροπολογίες ε, για τους τομιακούς κανονισμούς, τελικά τέθηκαν, μάλλον θέλετε, υπό την εξάρτηση του γενικού κανονισμού και τη ε, μοίρα που θα έχει. Δεν ξέρω, σε μοθοδολογικό επίπεδο, εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να κινούμαστε θεματικά και να μην κατακαιρματίζουμε ε, τι συναντήσει και τι συζητήσει ανά κανονισμό. Τώρα, επί τη ουσία. Ε, συμφωνώ πρώτα απ' όλα με τις ερωτήσεις και τους προβληματισμούς που εξέφρασαν οι σε ό,τι αφορά δηλαδή την χρήση των κονδυλίων για αυτόν τον μηχανισμό διασύνδεσης της Ευρώπης. Ε, να σε ρωτήσω το εξή. Πέρα από τη διαθεσιμότητά σας να συζητήσετε αυτό το θέμα κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Θα ήθελα μια πιο ξεκάθαρη θέση. Χθε εδώ ο Επίτροπος Κάλλας ενώπιον των δικών μας ενστάσεων και παρατηρήσεων μας μας απάντησε ξεκάθαρα, έξω από τα δόντια. Αυτή είναι η θέση μου, αυτή είναι η άποψή μου. Τέλος. Θα ήθελα λοιπόν να καταλάβω και από εσάς ποια είναι η δική σας θέση σε σχέση με τους κανόνες χρήσης των πόρων που θα ε, προέρθουν από το Ταμείο Συνοχής. Σε ό,τι αφορά τη θεματική συγκέντρωση, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Είναι πολύ σημαντικό να μην ανοίξουμε, αν θέλετε, αυτή τη συζήτηση και να μπαίνει ο καθένας με το δικό του θέμα. Ο καθένας και εγώ προσωπικά μπορώ να έχω προτιμήσεις, αλλά καλό είναι να εστιάσουμε προσοχή μας ε, στις θεματικές ενότητες που έχουν ήδη επιλεγεί. Πάντοτε λαμβάνοντας υπόψη είναι βεβαίως δική Ευρώπη 2020. Καλό όμως είναι να είμαστε πάντα ανοιχτοί να συζητούμε όλα τα θέματα και τι περιθώρια λιγμών υπάρχουν. Μιλάμε λοιπόν για θεματικές ενότητες που επιλέγονται με μια κάποια πολιτική διακριτική ευχέρεια, έτσι. Δηλαδή η Κομισιόν κάνει τις επιλογές. Εμείς στο Κοινοβούλιο κάνουμε κάποιες αντιπροτάσεις. Χρειάζεται λοιπόν να υπάρχει μια πολιτική, αν θέλετε, ευελιξία, ένα περιθώριο λιγμών, ώστε τελικά να καταλήξουμε στις θεματικές ενότητες που πιο πολύ ταιριάζουν στην Ευρώπη 2020. Είπατε επίσης ότι θα πρέπει να ενισχυθούν οι μηχανισμοί ελέγχου για να μειωθούν τα ποσοστά, ε, τα περιθώρια ασφάλματος. Ε, θα ήθελα να καταλάβω καλύτερα αυτοί οι ελεκτικοί μηχανισμοί κατά τη δική σας γνώση και κρίση όπως είδαμε και για την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, λοιπόν, κατά πόσο ελεκτικοί μηχανισμοί τελικά επηρεάζουν και συμβάλλουν στο ότι οι διαδικασίες είναι τελικά πολύ περίπλοκες και καταλήγουν ο τελικός δικαιούχος να λαμβάνει λιγότερα χρήματα. Πάρα πολύ γραφειοκρατία με άλλα λόγια, περίπλοκες διαδικασίες που κατά τη γνώμη μου τελικά επηρεάζει το τελικό αποτέλεσμα. Τέλος. Συμμετοχή των περιφερειών. Ορθά είπατε. Δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε την οργανωτική δομή που προβλέπεται σε κάθε κράτος μέλος. Άρα θα πρέπει εμείς να ερχόμαστε σε διάλογο με τον θεσμικό συνομιλητή όπως ορίζει το σύνταγμα της κάθε χώρας. Ορθό αυτό. Όμως, από την πλευρά μας, έχουμε και εμείς ένα σχεδιασμό που στοχεύει την περιφέρεια. Αυτός ο δικός μας σχεδιασμός τι σημαίνει συνεπάγεται ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας αναγνωρισμένος συνομιλητής που να εκπροσωπεί την περιφέρεια. Ακόμα και αν, αν θέλετε, το σύνταγμα της κάθε χώρας δεν προβλέπει έναν θεσμικό συνομιλητή σε επίπεδο περιφέρειας, πρέπει να υπάρχει. Είναι πολύ σημαντικό καθώς ε, μιλάμε για τον προγραμματισμό των περιφερειών για τη νέα περίοδο είναι καλό να ξεκαθαρίσουμε καλύτερα τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες ε, σε επίπεδο περιφερειών. Είμαι πεπισμένη ότι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πολλές χώρες, η Ιταλία μεταξύ αυτών, δυσκολίες λοιπόν να φέρουμε εις πέρας ε, τις υποχρεώσεις που έχουμε αναλάβει, οφείλεται σε ένα βαθμό στην ε, απουσία τέτοιων προσώπων στη φάση του σχεδιασμού. Γιατί θα πρέπει να υπάρχει ένα στρατηγικό σχεδιασμό αυτή εξ αρχή και θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει ο εκπρόσωπο των περιφερειών σε αυτή τη στρατηγική φάση του σχεδιασμού. Και τελικά, η αρχική στόχη να πρέπει να ελέγχουμε κατά πόσον επιτυχάνουν στο τέλο. Και βλέπουμε ότι η Ιταλία, για παράδειγμα, τι αντιμετωπίζει σήμερα. Πολλοί πόροι δεν έχουν απορροφηθεί από τι περιφέρειες του Νότου στην Ιταλία. Και Πού πάνε αυτά τα κονδύλια. Αναδιοχετεύονται από την κεντρική κυβέρνηση αλλού. Και δεν χρησιμοποιούνται αυτά τα κονδύλια για τις ε, νότιες περιφέρειες που τόσο μεγάλη ανάγκη έχουν, αλλά γενικά για το γενικό προπολογισμό, για να μην χαθούν τα κονδύλια. Είναι πολύ αρνητικό, δεν μπορεί κονδύλια που είχαν αρχικό δικαιούχο κάποιες συγκεκριμένες περιφέρειες του Νότου τελικά να καταλήγουν κάπου αλλού. Επίτροπε, έχουμε ακόμα τέσσερις ε, ομιλητές. Θέλετε να απαντήσετε στο τέλος? Ωραία. Βίκτορ Μπαστινάρου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε που ήρθατε εδώ σήμερα και για την ετοιμότητα και ευελιξία σας, ε, γιατί δεν ε, συμβαίνει πάντα αυτό με τους ε, συνομιλητές μας. Πρώτα απ' όλα, την προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο ο πρόεδρος ε, έκανε μία εξαιρετικά θετική ε, δήλωση και ομιλία για αυτό το ομοσπονδιακό σύστημα, το σωστό, αλλά μπορεί να λειτουργήσει μόνο με αλληλεγγύη. Ε, αλληλεγγύη έμπρακτη για τους Ευρωπαίους πολίτες. Δηλαδή αυτό, γι' αυτό απαιτείται ένας καλός αξιοπρεπής προπολογισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για την περιφερειακή πολιτική. Ιδάλλως ε, ο φτωχός ε, προπολογισμό μπορεί μόνο να υπονομεύσει αυτά τα προγράμματα. Από αυτή τη σκοπιά λοιπόν θα ήθελα να επαναλάβω την δραματική ανάγκη ε, να συνεργαστούν στενά η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο κατά τις διαπραγματεύσεις ε, του τριμερούς διαλόγου. Αυτό είναι θεμελιώδης σημασία. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που ήσασταν διατεθειμένος να το συζητήσετε και είστε τόσο θετικά διακείμενος ε, σε ό,τι αφορά τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις. Ένα θέμα μόνο. Τι συμβαίνει με την βελτίωση της διοικητικής ε, ικανότητας των κρατών μελών. Γιατί βλέπουμε τώρα ότι με μια τέτοια χαμηλή διοικητική ικανότητα ε, και το πιο καλό σχέδιο μπορεί να αποτύχει. Και τότε οι Ευρωπαίοι πολίτες ε, βεβαίως και δεν θα είναι φιλευρωπαϊστές. Προβλέπονται θετικές εξελίξεις με το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Εγώ είμαι πεπισμένος, μπορείτε όμως να το εξηγήσετε παραπέρα. Ε, χαίρομαι ιδιαίτερα με τις παρατηρήσεις σας για την ε, διευκόλυνση στην Ευρώπη. Και με το ανοιχτό πνεύμα της περιφερειακής πολιτικής και με την ε, δική σας προσωπική στήριξη μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα συμβασμό που θα συγκεράσει ε, την ε, τη DG Regio και την DG Move. Γιατί από, από δεύτερη προκύπτουν τα περισσότερα προβλήματα σήμερα. Είμαι πεπισμένο ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε και όλοι προς αυτήν την κατεύθυνση θα εργαστούμε. Τέλος. Θα ήθελα και στην Επιτροπή να ευχαριστήσω και εσά προσωπικά και γενικώ ε, την Επιτροπή για τον τρόπο με τον οποίο η Γενική Διεύθυνση ε, Περιφερειών ε, εργάζεται για την προετοιμασία των εκθέσεών μα και θεωρώ ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε συμβασμό μετά και την, με τις του Ιουλίου. Σίγουρα με το ίδιο πνεύμα θα συνεχίσουμε. Εδώ είμαστε όλοι πιστοί εταίροι. Ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής, κύριος Γκουτμάνης. Ευχαριστώ πολύ. Τι συμβαίνει με, με τους πόρους. Χωρίς πόρους ε, δεν μπορούμε να έχουμε ούτε καλούς κανονισμούς, ούτε καλή πολιτική. Θα γνωρίζετε ότι σε μια άτυπη ε, ε σύνοδος ε, στην Κύπρο κατέληξε σε απόλυτη καταστροφή η Κύπρος για πρώτη φορά έδειξε ότι η Κύπρος έχει επισήμως γράψει ότι τα, τα κονδύλια, οι πόροι για το MFF πρέπει να μειωθούν. Για την συνοχή είναι ήδη μικρότερα τα ποσά στην ε, πρόταση της Επιτροπής, ε, περίπου 6% αν εξαιρέσουμε το Connecting Europe που δεν είναι ε, πολιτική συνοχής. πολλά κράτη-μέλη επιμένουν σε περικοπές 100 δις, περίπου 5% του ε, συνόλου. Ο συνολικός προπολογισμός ε, στις δεσμεύσεις είναι 1-3. Και πού θα τα βρουν αυτά τα 100 δις, αν το πετύχουν. Δεν, είμαι, ε, δεν πιστεύω ότι όσοι θέλουν μια καλύτερη πολιτική συνοχή θα το δεχτούν. Αλλά πρέπει να βρεθεί ένας συμβιβασμός. και ο δεύτερος κίνδυνος ε, είναι για του χρόνου. Το Συμβούλιο έχει κάνει πρόταση για περικοπές 5 δις ε, στον προπολογισμό και πάλι περίπου 4%. Και σε ποιον τομέα στρέφονται όλοι για να κάνουν περικοπές, πρώτα απ' όλα στην ε, συνοχή. Και εγώ θέλω να τονίσω εδώ ότι το εργαλείο για όσους θέλουν να περικόψουν ε, στην ε, συνοχή είναι λανθασμένο. Πράγματι μένουν 200 δις που δεν έχουν, ε, δεν έχουν, πρέπει να ρευστοποιηθούν γιατί δεν έχουν απορροφηθεί. Όμω το 65% αφορά την ε, συνοχή. Το υπόλοιπο 35% είναι για άλλε γραμμέ του προπολογισμού. Έρευνα, ενέργεια, πολλά άλλα. Σχέδιο ανάκαμψη που, υπήρχε, που υπάρχει μέχρι το 2013. Αλλά κάπω πρέπει να λύσουμε αυτό το πρόβλημα και πρέπει να αναφερθείτε σε αυτό και εσεί. Γιατί είναι δύσκολο να απαντηθεί ένα ερώτημα. Σήμερα, αν δούμε τα δεδομένα. Ε, στο Ταμείο Συνοχής και στο Περιφερειακό Ταμείο υπάρχει 40% απορρόφηση από τα κράτη-μέλη. Στο Ταμείο Συνοχής είναι 45%. Δεν είναι κακό ω αποτέλεσμα. Το Ταμείο Κοινωνικής ε, Περιφερειακής Συνοχής ένα, ένα μικρό ποσοστό όπου υπάρχει μικρή απορρόφηση. Υπάρχουν βέβαια και τέσσερις χώρες που ξέρετε πολύ καλά ποιε είναι που τα πάνε πολύ άσχημα, 20-21% μεγάλες χώρες με πολλά χρήματα. Και αυτές οι χώρες τραβάνε όλους τους άλλους προς τα κάτω. Ε, δεν είμαι η δήμον. Αν ήμουν η Δήμων μάλλον στο Συμβούλιο, θα έλεγα, θα έλεγα όλον τον ε, όλον τον προπολογισμό και θα έλεγα ορίστε δεν, τα, δεν απορροφούνται τα κονδύλια, πρέπει να τα περικόψουμε. Όμως υπάρχουν μόνο καμιά δυο χώρες που τραβάνε τους υπόλοιπους κάτω. Αυτό πρέπει να καταστεί σαφές. Δυστυχώ, στην ομάδα των φιλελευθέρων εγώ είμαι εντελώ αντίθετος και οι χώρες από το Ταμείο Συνοχής θα είναι αντίθετοι αλλά στην ομάδα μου η πλειοψηφία ε, πρότεινε ε, τροπολογίες στις ομάδες για τον προπολογισμό 2013 ε, ώστε να τεθεί 30% ως αποθεματικό του Ταμείου Συνοχής και του Φραγκού Ταμείου μέχρι να ε, μας προτείνει νέο σχέδιο η Επιτροπή για καλύτερη απορρόφηση ακόμα και για την συμφωνία του επομένου MFF, το οποίο είναι ανοησίες. Αλλά αυτό δείχνει και τη στάση των Ευρωβουλευτών. Γι' αυτό κύριε Επίτροπε θα ήθελα να πω ότι άλλο να κάνουμε έναν καλό κανονισμό και σίγουρα ε, η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο καλά θα το κάνουν. Αυτό δεν είμαι σίγουρος για το Συμβούλιο, γιατί ήταν περίεργη λίγο η χθεσινή συνάντηση. Ούτε καν έχουν διαβάσει τι προτάσει μα αν με ρωτάτε, και τους ε, συμβιβασμού που προτείνουμε εγγράφω. Θα είναι δύσκολο λοιπόν. Πρώτα απ' όλα όμω πρέπει να υπερασπιστούμε του πόρου μα, γιατί πρόκειται για πόρους ε, που τη χάνουν συγχρηματοδότησης για το Connecting Europe, όχι τα υπόλοιπα. Είτε τα διαχειρίζονται τα κράτη-μέλη, είτε η Επιτροπή. Γι' αυτό σας παρακαλώ να το προσέξετε αυτό, γιατί θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα και για εσάς και για εμάς που είμαστε στην περιφερειακή πολιτική. Ευχαριστώ. Thank you, Petru Luhan. E, Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Εκτιμώ το ότι ο Επίτροπος ήρθε και μας παρουσίασε με τέτοιο λεπτομερή τρόπο την πρότασή του. Βεβαίως δεν καλύφθηκαν όλα τα σημεία και είχα την ευκαιρία ήδη να το ξαναπώ. Η κοινωνική συνοχή, η εδαφική συνοχή μιας ε, περιοχής μπορεί να διασφαλιστεί με πολύ συγκεκριμένους τρόπους. Το θέμα όμως της κοινωνικής ε, πολιτικής και της πολιτικής συνοχής είναι κάτι που δεν μπορούμε να το παρακάμψουμε. Χρειαζόμαστε καλές υποδομές. Χρειαζόμαστε δίκτυα. Χωρίς αυτά δεν υπάρχει ανάπτυξη. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό η χώρες να μπορέσουν να υποφεληθούν. Κύριε Επίτροπε, αυτά τα δέκα δις πώς θα κατανεμηθούν. Θα γίνει αυτό σε σχέση με τις ανάγκες των κρατών μελών, σε σχέση με την ποιότητα των ε, προγραμμάτων που θα υποβληθούν. Ένα μεγάλο ερωτηματικό έχουμε εδώ και θα ήθελα κάποιος να απαντήσει σε αυτή την ερώτηση. Δεύτερον, Κάτι που μπορεί να μας διευκολύνει, απλοποιώντας λίγο την ε, πολιτική συνοχής, είναι να υπάρξει μια διαφορετική αντιμετώπιση των μεγάλων σχεδίων που ξεπερνούν τα 15 εκατομμύρια ευρώ. Τι μέτρα θέλει να υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε η υποβολή των σχεδίων να απλοποιηθεί. Και εδώ πραγματικά Έχω κατά νου διάφορα σχέδια, διάφορα προγράμματα και η εμπειρία μέχρι τώρα μας δείχνει ότι η ανάπτυξη των κρατών μελών είναι τελείως διαφορετική. Από τη μία χώρα στην άλλη η κατάσταση διαφέρει πάρα πολύ. και ότι δεν είναι δυνατόν να αγνοήσουμε τις ε, λιγότερο αναπτύγμενες περιοχές ε, σε αυτήν την προσπάθεια. Τι μέτρα λοιπόν θέλετε να πάρετε για να απλοποιηθούν οι διαδικασίες. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, τις προάλλες στην Ολομέλεια ο πρόεδρος Μπαρόσο χρησιμοποίησε μία έκφραση που μας ικανοποίησε ιδιαίτερα εμάς εδώ στην Επιτροπή μας, ότι ο μελλοντικό ευρωπαϊκός προπολογισμό θα λαμβάνει υπόψη και θα προορίζεται για την εδαφική, οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και συνοχή. Ξέρετε, Έχουμε κάποιους προβληματισμούς όμως στην Επιτροπή μας σε ό,τι αφορά αυτό το μηχανισμό του συνδέοντος στην Ευρώπη, γιατί βλέπουμε ότι δεν εστιάζει στον οικονομικό, κοινωνικό και εδαφικό χαρακτήρα, αλλά επιλέγει ε, project με βάση την ποιότητα και την οριμότητα, χωρίς όμως να έχει βασικό γνώμονα την συνοχή κάτι που θεωρούμε ότι θα έπρεπε να συμβεί. Πρέπει λοιπόν να γίνουν κάποιε τροποποίησει. Επίση, θέλω να εκφράσω την ανησυχία μα σχετικά με την αλλαγή στον προγραμματισμό και την αναγκαιότητα συμμετοχή των περιφερειών και κατά τον προγραμματισμό και επιλογή των στρατηγικών σχεδίων. Εγώ έχουμε μια περιφέρεια που αυτή τη στιγμή εκτελεί κάποια κονδύλια που λόγω της κρίσης στη Γαλλικία, δεν μπορούμε να εκτελέσουμε, να χρησιμοποιήσουμε τα κονδύλια. Αυτό είναι μείζον για την διατήρηση και για την δημιουργία νέων εργασία. εργασίας. Και για να μην εγκαταλείπουν τις περιφέρειες μας οι νέοι, όπως συμβαίνει ήδη. Πώς μπορούμε λοιπόν να εγγυθούμε από τη μία την επιστροφή στην συνοχή, σε ό,τι αφορά το μηχανισμό συνήθω στην Ευρώπη. Και δεύτερον, πώ μπορούμε να έχουμε έναν μεγαλύτερο έλεγχο σε αυτέ τι αλλαγέ στον προγραμματισμό που γίνονται μέσα σε κάποια κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Πολύ σύντομα στο θέμα της διευκόλυνσης συνδέοντας την Ευρώπη. Η δική σας πρόταση εδώ θα ήταν πάρα πολύ σημαντική. Εμείς έχουμε υποβάλει με σαφήνεια το πώς βλέπουμε τα πράγματα. Εντάξει, δεν υπάρχει 100% υποστήριξη, υπάρχουν κάποιες ανησυχίες, το καταλαβαίνω. Γι' αυτό όμως και θα συνεχίσουμε την διαπραγμάτευση και θα πλησιάσουμε οι μεν δε. Γι' αυτό και σας καλώ και εσείς να καθορίσετε τη θέση σας δεν πρέπει να παραμένουμε με ασαφείς θέσεις. Πώς βλέπουμε εμείς τα πράγματα το ξέρετε. Από εδώ και πέρα θα πρέπει να δούμε και εσείς πώς αντιμετωπίζετε το θέμα. Το θέμα των πιο απομακρυσμένων περιοχών. Νομίζω ότι η προηγούμενη εβδομάδα μας έδειξε οι ανάγκες, οι προκλήσεις των διάφορων περιφερειών είναι τελείως διαφορετικές σε σχέση με το που βρίσκονται, αν είναι στο κέντρο, αν είναι απομακρυσμένες, αν είναι νησιά κτλ. κτλ. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε όλες αυτές τις ε, παραμέτρους. Και θα πρέπει επίσης να δούμε τι εννοούμε όταν μιλάμε για εξαιρέσεις. Ξέρετε ότι εμείς στην Επιτροπή πάντα είμαστε διστακτικοί όταν ακούμε για εξαιρεσει. Όταν όμως υπάρχουν ειδικέ δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπιστούν μόνο με ένα και συγκεκριμένο τρόπο, βεβαίως το παρελθόν μας έδειξε ότι είμαστε αρκετά ευέλικτοι και μπορούμε εδώ να αποφύγουμε περαιτέρω αποδυνάμωση κάποιων περιοχών, είτε επιδείνωση των δυσκολιών που ήδη αντιμετωπίζουν και το ίδιο πρέπει να κάνουμε βεβαίως και στον τομέα των μεταφορών, αλλά και σε άλλους τομείς. Ένα νησί, παραδείγματο χάρη, μπορεί να αντιμετωπιστεί τελείως διαφορετικά και βεβαίως διαφορετικά αντιμετωπίζεται ένα νησί που είναι απομονωμένο κάπου, είτε μια ομάδα νησιών, Κανάριες νήσους, η Μαρτινίκα. Εν πάση περιπτώσει έχουμε εδώ κατά νου το γεγονός ότι βεβαίως υπάρχουν τα ειδικά ενδιαφέροντα και συμφέροντα κάποιων περιοχών που θα πρέπει να ειδωθούν ολοκληρωμένα στο πλαίσιο της γενικότερης πολιτικής μας. Επαναλαμβάνω ότι εμείς κάναμε τις προτάσεις μας, δώσαμε και κάποιους λόγους για τους οποίους οδηγηθήκαμε σε αυτές τις προτάσεις, αλλά από εδώ και πέρα εσείς πρέπει να αντιδράσετε. Και την προηγούμενη εβδομάδα εγώ είπα σε όλους τους εκπροσώπους κάποιων περιοχών περιφερειών ότι και τα κράτη-μέλη έχουν κάποιες υποχρεώσεις, κάποιες αρμοδιότητες, τις οποίες καλούνται να ολοκληρώσουν. Υπάρχει μια αλυσίδα, αν θέλετε, υποχρεώσεων και επιπέδων. Το ευρωπαϊκό επίπεδο, το εθνικό επίπεδο, οι περιφέρειες, οι τοπικές αρχές. Και θα πρέπει όλα αυτά να συντονιστούν. Μιλήσατε για τις υποδομές, ναι. Βεβαίως, χωρίς να πέσουμε σε αντιφάσεις και εδώ θα πρέπει να δείξουμε μια σχετική ευελιξία όσον αφορά τους ορισμούς. Γιατί καταλαβαίνετε ότι ένας πάρα πολύ άκαμπτος ορισμός μπορεί να περιορίσει σημαντικά τις δυνατότητες χρηματοδότησης και επενδύσεων. Δεν θέλω τώρα να μπω σε συγκεκριμένες διευκρινήσεις, αλλά θα ήθελα πραγματικά να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα γιατί πολλές περιφέρειες, πολλές περιοχές που έχουν συγκεκριμένες ανάγκες έχουν ήδη αναλάβει πρωτοβουλίες. Παραδείγματο χάρη χρηματοδότηση ενός οδικού δικτύου, μια πολύ συγκεκριμένη αν θέλετε, προτεραιότητα που έχουμε θέσει στη στρατηγική 2020 για την Ευρώπη και εδώ θα πρέπει όλοι να παίξουν το ρόλο τους. Τώρα, για τον έλεγχο. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπατε. Το είπα και εγώ όμω στα εισαγωγικά μου σχόλια. Σύμφωνα με αυτά που εγώ πρεσβεύω και οι πραγματογνώμονες της Επιτροπής συμφωνούν, το θέμα δεν είναι η επιπλέον έλεγχη. Ο στόχος μας είναι κοινό. Θέλουμε να παραμείνει σταθερός ο αριθμός των ελέγχων. Ξέρετε ότι το ελεγκτικό συνέδριο στις αναλύσεις του φτάνει πάντα στα ίδια συμπεράσματα, σε γενικές γραμμές. Ο έλεγχος που γίνεται καλύπτει ικανοποιητικά, πάντα υπάρχουν εξαιρέσεις, αλλά ικανοποιητικά το έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, ίσως σε κάποια σημεία χρειάζεται λίγο παραπάνω προσπάθεια, αλλά δεν νομίζω ότι ο επιπλέον αριθμός ελέγχων είναι εδώ το ζητούμενο. Εταιρικές σχέσεις, εταιρικές συμβάσεις. Αυτά που είπατε είναι 100% ορθά. Τώρα το θέμα ίσως είναι η διατύπωση των προτάσεών μας, οι οποίες πολλές φορές μπορεί να οδηγήσουν σε κάποιες παρερμηνίες. Πώς βλέπουμε εμείς το θέμα αυτό. Και ελπίζω να το καταλαβαίνετε και εσείς με τον ίδιο τρόπο. Η σύναψη αυτών των συμβάσεων των εταιρικών θα πρέπει να γίνεται ταυτόχρονα με την υποβολή των προγραμμάτων. Βεβαίως, οι διαπραγματεύσεις γίνονται σε διάφορες ε, διαδοχικές φάσεις. Τελικά όμως, τελικά θα πρέπει τα προγράμματα αυτά να οδηγούν σε αυτές τις ε, εταιρικές σχέσεις και το ξεκίνημα, αν θέλετε, της υλοποίησης να γίνεται ταυτόχρονα με την σύναψη. Ε, με κάποιο τρόπο δηλαδή θα πρέπει εδώ λίγο να εναρμονιστούν οι διαδικασίες. Όσον αφορά τώρα τις διοικητικέ ε, δυνατότητες, εδώ πρέπει να βελτιωθεί και ποσοτικά αλλά και κυρίως ποιοτικά. Σε κάποιες χώρες θα πρέπει να βελτιωθεί το νομικό, το νομοθετικό πλαίσιο. Πολλές φορές υπάρχει σύγχυση μεταξύ των επιπέδων εθνικό, περιφερειακό, τοπικό. Δεν υπάρχει μία και μοναδική συνταγή βεβαίως εδώ. Καταλαβαίνω ότι πολλές φορές σε εθνικό επίπεδο υπάρχουν κάποια εμπόδια. Εγώ ήμουν υπουργό, ξέρω πως οι διάφορες διαδοχικές διοικητικές αρχές μπορεί να κατανείμουν με δύσκολο τρόπο τις διάφορες αρμοδιότητες, αλλά εν πάση περιπτώσει εδώ θα πρέπει να αποφασιστεί ποιο είναι το αρμόδιο επίπεδο και να μην αλλάζει συνέχεια. Νομίζω λοιπόν ότι στα περισσότερα που άκουσα από εσά μπορώ να συμφωνήσω 100%. Η ερώτηση τι θα γίνει αν δεν συμφωνήσουμε για το δημοσιονομικό πλαίσιο. Δεν το είπατε τόσο ξεκάθαρα, αλλά οι ανησυχίες σας ουσιαστικά ε, αυτό με οδήγησε να καταλάβω. Μα αυτό θα είναι κάτι που πραγματικά δεν ξέρω αν μπορούμε να το φανταστούμε. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή χρειάζεται πολύ συγκεκριμένα μηνύματα, αξιοπιστία, και χρήματα τα οποία με μια ασφάλεια, με μια σιγουριά θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Η ροή των κονδυλίων, όπως είπατε, θα πρέπει να διασφαλιστεί. Και πιστεύω θα υπάρξει εδώ συμφωνία. Βέβαια, εντάσεις πάντα υπάρχουν από τις διαπραγματεύσεις στο Συμβούλιο. Παρατηρούμε και αυτό είναι σημαντικό αυτό που έγινε στην Κύπρο, ότι η Ιταλία, παραδείγματος χάρη, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, που ανήκουν στην ομάδα των φίλων της πολιτικής της συνοχής, αναγνωρίζουν παρόλα αυτά κάποιες ανάγκες. Γι' αυτό και έγινε μια έκκληση, την οποία εγώ επαναλαμβάνω εδώ, για περισσότερες κοινέ θέσεις. Μην πιστεύετε ότι οι διμερείς συμφωνίες θα μπορέσουν να μας γλιτώσουν από μια κοινή προσπάθεια να πλησιάσουμε ή μεν τους δε. Η κάθε δημοσιονομική, αν θέλετε, συζήτηση μπορεί να επηρεάσει, να πλήξει όλη την πολιτική συνοχής. Αλλά θα πρέπει πραγματικά να υπάρξει ένας επικοδομητικός διάλογος και μια εξισορροπημένη προσέγγιση μεταξύ όλων των στόχων, μεταξύ των περισσότερων και λιγότερων αναπτυγμένων περιοχών της Ευρώπης και θα πρέπει ο στόχος μας να είναι πάντα ευρωπαϊκός. Δεν μπορούμε να στοχεύουμε μόνο τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες βέβαια. Γιατί τι θα γίνει στην επόμενη θητεία ή στην παραεπόμενη θητεία ή σε δύο ή τρεις θητείες δεν θα υπάρχουν πλέον διαρθρωτικά ταμεία. Θα πρέπει να δούμε πώς εποφελούνται οι περιοχές από τα χρήματα που λαμβάνουν. Έχετε δίκιο σε αυτό. Η περιφερειακή πολιτική είναι η καρδιά του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Και σκοπός μας είναι εδώ να βελτιώσουμε την υλοποίηση αυτής της πολιτικής. Να δημιουργήσουμε κανονισμούς και σαν πολιτικός που δεσμεύομαι στην πολιτική των περιφερειών, θα ήθελα πραγματικά να ζητήσω και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από τα κράτη-μέλη αυτό το μήνυμα να συνεχίσει να είναι ζωντανό οι διαπραγματεύσεις φυσικά θα συνεχιστούν και ελπίζουμε με θετικό αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνεργασία. Ευχαριστώ και εξ ονόματος των συνεργατών μου και θα ήθελα να σας επαναλάβω ότι είμαι στη διάθεσή σας γιατί σκοπός όλων μας είναι τελικά να είναι καλύτερο το μέλλον της Ευρώπης. Σας ευχαριστώ. Thank you, Commissioner. We have not clearly... Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Είπατε, είχατε τον τελευταίο λόγο, πράγματι χρειάζεστε την ε, βοήθειά μας για να μπορέσει να καταλήξει στην πλέον ε, καλύτερη λύση για το CF και πράγματι αυτό είναι καθήκον του Κοινοβουλίου. Λοιπόν, καλώ όλους τους συναδέλφους εξ ονόματος της ε, Ρίκα και της Μαρίς Τερέζ να στρατηθούμε εδώ έξω. Και ο Επίτροπος θα μπορούσε να μείνει λίγο μαζί μας να τοποθετηθεί για αυτό το θέμα της σημασίας της συνεργασίας στην Ευρώπη. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε στις 3.